So, liebe Kolleginnen Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ βγάλτε τις κάρτες σας για τις ψηφοφορίες. Einführen und dann gleich losgehen. Για να ψηφίσουμε. Ετοιμάστε τα μηχανήματα. Αλλάξαμε λίγο την ημερήσια διάταξη και βάλαμε πρώτα την ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 88 απαιτήσει οικολογικού σχεδιασμού των ε, βραστήρων και ε, δεξαμενών αποθήκευσης του νερού. και των θερμοσυφώνων. Το 9 παραμένει και μετά έχουμε το 10. Νέα εκβιομηχάνηση της Ευρώπης για την παραγωγή την προαγωγή συγγνώμη, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας. Και μετά έγινε μια αλλαγή. Θα ψηφίσουμε μετά το 12 το 11 πρώτα τα φθοριούχα αέρια και μετά το backloading. Για να ξέρετε όλοι με ποια σειρά ψηφίζουμε. Λοιπόν, το 12 έχει αντιστραφεί με το 11. Αυτή είναι η αλλαγή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την ένσταση πρώτα, σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2. Άρχεται η ψηφοφορία και είναι ηλεκτρονική, παρακαλώ. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Μία ψήφος υπέρ και 51 κατά. Only Karl Schlüter is in favor. Ο Καρλ Σλούτερ υπερψήφισε. I thought we were voting fluorinated gases. Sorry. Ε, νόμιζα ότι ψηφίζαμε τα φθοριούχα. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα. Με τα μηχανήματα. Ο κύριος Λούτερ επιθυμεί να αλλάξει την ψήφο του να τη διορθώσει. Κατά λάθο υπερψήφισε. Κατά ήταν κι αυτός. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η δική μου έκθεση. Ψηφίζουμε το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου για το σημείο 9. Είναι μία και μοναδική πάλι ε, ψηφοφορία. ηλεκτρονική αρχίζει τώρα. Η τροποποίηση των αντιστοίχων οδικιών. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 54 υπέρ, 2 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν για η πρόταση αυτή. Προηγούμενη περίφθη. Συνεχίζουμε. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Σιμάνσκι. Νέα εκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Και αρχίζουμε. Τροπολογία παριθμών 19 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την 20. Αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ παρακαλώ. Δύο και τώρα. Υπεράριθμος είπα, όχι λιγότερος. Α, τώρα είμαστε εντάξει πέρας. 31 υπέρ, 27 κατά και μία αποχή. Δεν κρίνεται. Η τροπολογία 21 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 21 ηλεκτρονικά και πάλι αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Ξεκολουθεί να είναι ένας υπεράριθμος. Θα είχε κανείς την καλοσύνη από το ΕΛΚ να βγάλει την κάρτα του, σας παρακαλώ. Εγκρίνεται. 31, 29, μία αποχή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. 23 χρειάζεται ηλεκτρονικό έλεγχο. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πες. Εγκρίνεται. 24 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 37 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 25 είπε. Κατά. Και αυτή χρειάζεται ηλεκτρονικό έλεγχο, δεν ψηφίζεται. 25 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι, πέρας. Καλά. Εντάξει. Εγκρίθηκε σαφώς. 26 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την ενοποιημένη Consolidated 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η συνδυασμένη. 28 κατά τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά Αποχές επίσης εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Consolidated 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41. Κατά τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. πίπτη 42 και ερχόμαστε στην ενοποιημένη 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 3 Επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 57 Επέ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές όμως. Ξανά 57 Επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα 58 Επέ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 58 παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Περάσα. Εγκρίνεται. κρίνεται. δύο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε και πάμε στην 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Τσεκ φωνάζουν από κάτω. Ωραία. Έλεγχος για την 71 ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 72 επέ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 επέ Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. 77, 78 και 79 μαζί, είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 83 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Έλεγχος για την 83 παρακαλώ τώρα ηλεκτρονικά. Αν ψηφίσατε όλοι, λίγη ψηφοφορία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δύο τώρα παραπάνω είναι. Λοιπόν, τώρα είμαστε εντάξει. Εγκρίνεται. 84 είπε. Αποχέ. Άποχες. Ε, μόνο 10% σηκώνουν χέρια, οπότε ηλεκτρονικά τώρα. 84 έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται. 85 και 86 μαζί. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συνεχίζουμε στην 91. Είμαστε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92. Κατά τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 92. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 93 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 94 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές όμως 99 ηλεκτρονική επαλήθευση ψήφισατε όλοι το ΕΛΚ παραμένουν δύο παραπάνω Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. 101 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε 103 κατά τμήματα. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. 103 σκέτη υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Εδώ είναι το χωριστή. 104 αλλά καταπίπτει όπως και 105 και 106. 107 υπέρ. Σε 107. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 111 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 είπέ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 Ich weiß nicht, sollen wir eine kurze Sitzungsunterbrechung machen, oder? Θέλετε μικρή διακοπή τη συνεδρίαση για να συνεχίσετε τι ιδιωτικέ συνομιλίε. ενοχλείτε. Ε, ε, αυτά είπε. κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. αιτιολογική σκέψη α, 8, 9, 10, τροπολογία μαζί. Είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 11 και ερχόμαστε στη 13 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 είπε. Το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Τι ψηφίζουμε, 14 το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά. 12 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ερχόμαστε τώρα στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα ψηφίσατε όλοι πέρασε 54 υπέρ, 7 κατά, 5 εποχές. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή μας. Συνεχίζουμε. Τώρα είναι τα φθοριωμένα αέρια. Το 12 δηλαδή που έχουμε προτάξει. Yes, please. So, jetzt starten wir die Abstimmung zu den F-Gasen. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Η πρώτη ενοποιημένη τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Μάλιστα. Το ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Στα φθοριούχα ή φθοριωμένα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μα το είπαμε το πρωί στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, αλλάξαμε τη σειρά. Λοιπόν, άλλη απόπειρα καινούργια. Αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη το πρωί. Το διευκρίνησα στην αρχή της συνεδρίασης τώρα. Ψηφίζουμε την έκθεση ΕΚΧΑΟ, τα φθοριούχα αέρια και ελπίζω να έχετε και το σωστό κατάλογο ψηφοφορίας και να ξέρετε όλοι τι ψηφίζετε. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, Consolidated 1 στα φθοριούχα αέρια ηλεκτρονικά ζητήθηκε να ψηφίσουμε, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Το ΕΚ γίναν τρεις παραπάνω, ωραία. Zwei. Δύο παραπάνω ακόμα από το ΕΛΚ. Τι να κάνουμε, να διακόψουμε τις συνεδρίες. Ένας, άντε λίγο ακόμα. Παραμένει ένας υπεράριθμος βουλευτής του ΕΛΚ, ο οποίος ψηφίζει. Ρίχαρτ Σέμπερ. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ζητώ μικρή διακοπή της συνεδρίας για να κανονίσουμε ποιοι θα ψηφίζουν. Πόση ώρα θες, Ρίχαρτ, ε, τρία λεπτά το πολύ. So, die Sitzung... Εντάξει, επανάληψη συνεδρίασης. Αλλιώς θα αποφασίσω εγώ. Θα σας διαβάσω ποιοι είναι μέλη και ποιοι αναπληρωτές και να δείτε πώς θα το λύσουμε. Θέλετε να σας αναγνώσω τα ονόματα, τακτικά μέλη και αναπληρωματικά. Γνωρίζουμε και νέους συναδέλφους έτσι, ξέρετε. Ich glaube, jetzt wir Λοιπόν, τώρα είμαστε νομίζω εντάξει. Θα προσπαθήσω ξανά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Συνέκθεση για τα φθοριούχα αέρια, την ενοποιημένη τροπολογία 1, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τι θα γίνει με αυτό το ΕΛΚ, δύο είστε παραπάνω, τι θα γίνει παιδιά, θα ψηφίσουμε σήμερα. Soll ich noch mal die Namen vorlesen? Να σας διαβάσω τα ονόματα των μελών και των αναπληρωτών. Θέλετε να το κάνουμε έξι. Να, κάνουμε, να πάρουμε παρουσίες. Ποιος είναι τακτικό μέλος, ποιο αναπληρωματικό. Τόσο δύσκολο είναι. Δεν μπορείτε να το, χωρίσετε, να το αποφασίσετε. Λοιπόν, τρίτη απόπειρα. Τρίτη. τρίτη. Φθοριωμένα, area consolidated, τροπολογία επαριθμών 1, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 42 υπέρ, 21 κατά, καμία εποχή. Συνεχίζουμε. Η τροπολογία 86. Υπέρ. Κατά. Άποχες δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 86 ηλεκτρονικά. 86 ηλεκτρονικά Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 89 ψήφιπε. Κατά. Αποχές. Και εδώ χρειάζεται ηλεκτρονικό έλεγχο. Για την 89 παρακαλώ ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. «33 υπέρ 29 κατά εγκρίνεται». Συνεχίζουμε, αμπλόκ τώρα. 87, τραν 8, 90, τραν 9, 91 και τραν 10. Υπέρ. Είναι και της Επιτροπής Μεταφορών μερικές. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 93 ε, και 311. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92. Ορίστε. Συνεχίζουμε 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Consolidated 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 101 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Ή 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η 107 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται αν δεν απατώμε, αλλά θα το ελέγξουμε. 107 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 108 είπε Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Τις 108 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 είπε, κατά, αποχέση γκρίνεται, 111 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 είπε. Κατά. Να πω και έτσι εγκρίνεται. Η 12 των μεταφορών είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά στην ελέγξουμε. 116 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τσεκ. Έλεγχος λοιπόν για την 117. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Ε, κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 120-122 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι σαφές όμως 125 ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 και 129 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. Ωραία. Και τις δύο μαζί. 127-129 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεν κρίνεται σαφέστατα. Συγχαρητήρια. 128 και 13 καταπίπτουν, 130 τώρα υπέρ δεν έχει αποσυρθεί αυτή. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135. Το πρώτο τμήμα. Χωρίς την ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Ε, απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 130, όχι, 133 ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα. Ψήφισατε όλοι. Πέρα. 35 κατά 32 υπέρ 134 υπέρ. Κατά. εποχές έγινε. 34 και 15 δεν ψηφίζονται, είναι γλωσσικές. 10 και 136 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνονται. 11, 137, 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 140 ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ψηφίσατε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με διαφορά. 143 πέ. 143. Εκατά. Αποχές απορρίπτεται. 142 πέ. Κατά. Αποχές Δεν είναι σαφές πάλι. 142 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην ενοποιημένη παριθμόν 6 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και γυρνάμε σελίδα 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 Επέ. κατά αποχές εγκρίνεται. 162 Επέ. κατά αποχές εγκρίνεται. 165 Επέ. κατά αποχές εγκρίνεται. Και καταπίπτουν μερικές και πάμε στην 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και κάνουμε ένα άλμα τώρα με χαρά Πάμε στη σελίδα 14 παρακαλώ, 217 ανθρωπολογία. τα βρήκατε, σελίδα 14, 17 ε, ε, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε. 216 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται, 218 υπέρ. Κατά, Αποχές εγκρίνεται. 220, τραν 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 221 ε, και τραν 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές έλεγχος. Τη 222 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 224 είπε. Τι έγινε, 223. Τι ε, λάθος έκανα. 223 είπε Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 224 Πέ. κατά άποχες απορρίπτεται. Τώρα πάμε στη συμβιβαστική υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και άλλο άλμα τώρα. Ερχόμαστε στη σελίδα 19, ενοποιημένη 4, κάτω-κάτω. Το βρήκαμε. Ωραία, συνεχίζουμε υπέρ. Κατά, άποχες, εγκρίνεται. Άλλο άλμα, ενδιασμένη 3, σελίδα 21, υπέρ. Κατά, άποχες, εγκρίνεται. 285 τώρα είπε. Στη σελίδα 22. Υπέρ της 285. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση της 285. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 284 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τσεκ. Ωραία. Για τη 284 λοιπόν επαλήθευση τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ορίστε. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ πολύ Μπάς. 34 34 πίπτη 2,96 είπε. Όχι, 2,92 διορθώνει ο πρόεδρος, συγγνώμη. 292 είπε. Κατά, άποχες, απορρίπτεται. 2,93 υπέ, Κατά, άποχες, εγκρίνεται. Νομίζω. 2,94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και 36 πε κατά αποχές εγκρίνεται. 95 πε κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Δύο ταυτόσημες. Τραν 39 ε, υπέρ και 307-308 κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο 309 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 310 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 311 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 313 υπέρ Έλεγχος. 3.13 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 3.14 και τραν 40 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.15 και 3.41 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.16 και 3.42 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτω. Πάμε παρακάτω στη σελίδα, μια στιγμή να σας πω. «35 παρακαλώ». Τι έκπληξε αυτή. Στην 4.13 είμαστε. Υπέρ. Σελίδα 35 στο δικό μου κατάλογο είναι η τροπολογία 413. Το βρήκατε? Ωραία. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 414 και 345 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 415 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα block vote διάφορους τοπολογίες της Επιτροπής Μεταφορών, 46 με 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψεται 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψεται 59 υπέ. κατά αποχές αλλά έχουμε ηλεκτρονικά την 59 ε, Ψηφίσατε όλοι, παιδες. 39 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε 60 και 31. Υπέρ, είναι μα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 1 και 62 και ερχόμαστε 64 ψήφι υπέρ. Κατά. άποχέ 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. 66 υπέρ. Α, και η τραν 3 μαζί. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη σελίδα 38. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. Τσεκ. Εντάξει, ας το ελέγξουμε. Την 77. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Τι έγινε. Πάλι το ΕΛΚ έχει ένα παραπάνω. 77 ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Το ΕΛΚ έχει έναν υπεράριθμο ξανά. Τώρα, λίγη ψηφοφορία. 44 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται λοιπόν. Συνεχίζουμε. Η τροπολογία υπάρχει λοιπόν 6 ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τσεκ. Καλά. Ε, για καλό και για κόκο δεν είμαι σίγουρος, ας το αλλάξουμε. Ψήφισατε όλοι. Πέρασα. 35 υπέρ, 33 κατά. Εντρίνεται. 81 και 35 υπέρ. Κατά. Άποχες Εντρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα φτάσαμε ήδη στην τελική ψηφοφορία. η ηλεκτρονική πρώτα, καταρχήν. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 48 υπέρ, 19 κατά και μία αποχή. Τώρα έχουμε και άλλη ηλεκτρονική, το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Ψηφίσατε. Πέρας. 47 υπέρ 18 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Μπάς Αικχάουτ. dann frage Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 70 του κανονισμού. Βλέπω να συμφωνείτε. Οπότε χρειαζόμαστε 35 ψήφους, αλλά τώρα έχουμε απαρτία σήμερα, είμαστε όλοι εδώ. Κανονικά θα τις βρούμε και Ε, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για τη χορήγηση εντολής. Διαπραγματευτικής ψηφίσατε όλοι. Περά. 49 υπέρ, 16 κατά. Σαφέστατη εντολή, χαρακτήρια κύριε Σιγητά. Bitte noch nicht den Saal verlassen. Μην φύγετε ακόμα, έχουμε άλλη μία. Μην διστάσετε να συνεχίσετε να ψηφίζετε. Nie, nie, to jest coś innego, to jest zupełnie coś Λοιπόν, πριν μπούμε στη ψηφοφορία για το λεγόμενο backloading, το βαρές χρονοδιάγραμμα, να σας πω κάτι διαδικαστικά τώρα για την ψηφοφορία. Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 157 του κανονισμού, οι τροπολογίες 23, 36, 54 και 62 δεν είναι παραδεκτές. Έτσι. Α, έχουμε και τηλεόραση. ΑΡΤ, ε, ε, ΤΒΠ, πολωνική τηλεόραση, και γερμανική ΑΡΤ και Europe Satellite. Λοιπόν, αυτές οι τροπολογίες που σας είπα δεν είναι παραδεκτές βάσει κανονισμού. Το λόγο ζήτησε η κυρία Κόρχολα, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να παρακαλέσω να ψηφίσουμε για την τροπολογία 21 γιατί είχα ψηφίσει κατά της διαδικασίας ε, έγκρισης σε πρώτη ανάγνωση στην Επιτροπή αυτή. Νόμιζα ότι θα έπρεπε το σώμα να έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί. Όχι μόνο η πολιτική μου ομάδα. Βεβαίως το αποτέλεσμα της Επιτροπής ΕΝΒΗ δεν θα αντικατοπτρίζει πλέον την βούληση ολόκληρου του σώματος. Το αποτέλεσμα στην ψηφοφορία του Απριλίου στην Ολομέλεια αυτό απέδειξε. Τώρα ψηφίζουμε για το ίδιο πράγμα και ως και εισηγήτρια για την ομάδα μου θέλω να δηλώσω ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί το ΕΛ και το τι θα γίνει στην Ολομέλεια με αυτή την ψηφοφορία. Πρέπει να υποθεί πριν ψηφίσουμε, ώστε κανεί να μην κατηγορήσει τα μέλη τη ομάδα μου εκ των υστέρων. Ω σκιώδη εισηγήτρια, πρέπει να πω ότι συνολικά η ομάδα δεν έχει αλλάξει. τη θέση να απορριφθεί το backloading όπως προτείνεται. Αυτή είναι η δική μου θέση ω εισηγήτρια και είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Κυρία συνάδελφε, βάση... Α, όχι, ο Ρίχαρτ Τσέμπερ πρώτα. Θα ήθελα να πω ότι η Συναδελφο Κόρχολα δεν ομιλεί εξ ονόματος ε, της ομάδας. Εχθές επίσημα άρχισε μία ε, συνεδρίαση, ε, ψηφίσαμε και την άλλη εβδομάδα θα δούμε τι άποψη θα έχει το σύνολο της πολιτικής ομάδας και πέρα από την ομάδα εργασίας και αυτή είναι η θέση μας ως ομάδα. Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 195 μπορεί να ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία εφόσον συμφωνήσουν 18 συνάδελφοι και εγερθούν, αλλιώς δεν θα υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ, σηκωθείτε δηλαδή. Κυρία Κόρχολα, μόνο είστε. Πρέπει να εγερθούν, παρακαλώ να σηκωθούν οι συνάδελφοι που ζητούν να γίνει αυτό. Είναι πάνω από 18. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε και ονομαστικά. Είναι πάνω από 18 οι συνάδελφοι. Ε, τεχνικά χρειάζεται κάποια ρύθμιση αυτό. Λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει τώρα η ονομαστική για την τροπολογία αριθμών 21 και 22. Όχι, διορθώνει ο 21 μόνο μέχρι την αιτιολογική σκέψη 3. Τρει από το ΕΛΚ και υπεράριθμοι. Τι έγινε τα αρχίδια, θα ξαναρχίσουμε. Δύο τώρα. Ένα Ένας, αντίστροφη μέτρηση. Τώρα είμαστε εντάξει, το βρήκαμε. Λοιπόν, τώρα αρχίζει η ηλεκτρονική όσο και ονομαστική ψηφοφορία. Πάλι ένας από το ΕΛΚ παραπάνω. Τι κάνουμε. Παιδιά, α, τώρα οι φιλελεύθεροι, ωραία. Ένας παραπάνω. Και από το ΕΛΚ ακόμα περισσεύει ένας. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ένας υπεράριθμος. Wir können die Abstimmung nicht durchführen. Δεν μπορούμε να κάνουμε ψηφοφορία όταν ψηφίζουν υπερβολικά πολλοί συνάδελφοι. Ε, το ΕΛΚ αντί να ε, φερεί προσθέτει. Τώρα είναι δύο παραπάνω. Ένα zu viel. Ένας ακόμα. Es ist immer noch ein Mitglied der EVP. Παραμένει ένας του ΕΛΚ υπεράριθμος, πώς να σας το πω. 24 haben Sie. Έχετε 24 μέλη αν δεν έχετε καταλάβει. Συμφωνήστε ποιος αναπληρωτής ε, θα ψηφίσει ή από τους νέους που βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου στην Επιτροπή. Ich weiß, Sie haben eine polnische Έχουμε εδώ μια Πολωνή συνάδελφο, το ξέρω. So, jetzt. Βρήκαμε. Εντάξει. Λοιπόν, πέρα τη ψηφοφορία. 44 κατά 23 υπέρ και μία αποχή. Haben wir Ja, den Ausdruck haben wir, so dass es λοιπόν, το τυπώσαμε κιόλα και έχουμε και στοιχεία και επιστήρια Ποιο ψήφισε τι και συνεχίζουμε. Ε, με την ενοποιημένη τοπολογία υπερφών 1, πάλι ηλεκτρονικά αμέσω, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Consolidated 1. 38 υπέρ 27 κατά και μία εποχή Ούτως και εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Η τροπολογία παριθμών 70, 24 μέχρι και 50. Μαζί όλες αυτές, στη σελίδα 3. Ηλεκτρονικά, γιατί είναι τόσο ωραίο και μας αρέσει, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 33 υπέ 33 κατά. ψηφία απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Στην 71. Ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τσεκ Άρα έχουμε την 26 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε. Τέλος. Απορρίπτεται. 36 κατά, 31 υπέρ. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 δεν ψηφίζεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 38 ψήφισατε όλοι πέρας 39 υπέρ 28 κατά εγκρίνεται η 38 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ενωποιημένοι δύο. ηλεκτρονικά αμέσω. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 47 υπέρ 19 κατά και μία αποχή. Η 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα η 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας την ελέγξουμε καλύτερα όμως την 52. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά ας την ελέγξουμε καλύτερα. ψήφισα τέλεια. Πέρας. 33 υπέρ, 35 κατά. Απορρίπτεται. Δύσκολα. Και η 46 τώρα υπέρ. αποχές απορρίπτεται 47 είπε; κατά αποχές απορρίπτεται 49 τσεκ καλά ελέγχουμε τη 47 ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίες απορρίπτεται ισοψηφία 33-33 συνεχίζουμε 49 είπε. κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος πάλι για την 49 ψηφίσατε όλοι πέρα εγκρίνεται 37 υπέρ 25 κατά και δύο αποχές 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 56. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. 25 υπέρ, 42 κατά. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος της ψηφοφορίας. Τι έγινε, 59, δεν την ψηφίσαμε. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, πολύ ωραία. Ψηφίζουμε. Την 59 ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 35-33. Λοιπόν, τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Δεν ήταν εύκολη η ιστορία αυτή με την έκθεση. Και τώρα, χωρίς τροπολογίες, πάει αμέσως στην Ολομέλεια. Και στην αμέσως επόμενη σύνοδο θα το ψηφίσουμε το πράγμα για να τελειώνει η υπόθεση. Σας ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό σας και το πνεύμα προθυμίας που δείξατε για συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Hans Gross Meine Damen und Herren, Λοιπόν, αν ε, επανέλθει σιγά σιγά η ηρεμία θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, να πάτε στο καλό, αλλά ησύχω για να μπορέσουν οι υπόλοιποι να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση. Ε. Ερχόμαστε στο σημείο 13 τώρα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για την ησυχία. Τροποποίηση τη οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και της οδηγίας σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Παρένθεση. Έμεση αλλαγή ε, της χρήση γη. Κλείνει παρένθεση. Η συγκήτρια είναι η κυρία Κορίν Λεπάς και έχει αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε σε ένα θέμα κάπως πιο θερμό από το backloading, λιγότερο θερμό από το backloading λοιπόν, αλλά από γύρει πολλά προβλήματα. Υπάρχουν ε, εκατοντάδες τροπολογίες για την έκθεση που συνέταξα και θα προσπαθήσω σήμερα να σας δώσω κάποιες γενικές ε, γραμμές συμβιβασμού. Περί τίνος πρόκειται έχουμε να κάνουμε με δύο κείμενα. Το ένα ως προς την ποιότητα των καυσίμων του 2009, το άλλο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα κείμενο που προβλέπει ως το 2020 10% στις μεταφορές τη ενέργεια που καταναλώνεται στι μεταφορέ να καλύπτεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Δεν είπε γιατί καύσιμα πρόκειται, αλλά ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Το κείμενο αυτό έτυχε πολλών διαφορετικών ερμηνεών, ιδίω από όσου είχαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και δεν μπορούμε βεβαίω να του το ε, καταλογίσουμε αυτό, για το στόχο του 10% των βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς όπως λέγονται το 2020. Βιοκαύσιμα λοιπόν τα οποία παρασκευάζονται από εδόδημα θετικά προϊόντα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, το βιοντίζελ το οποίο έχει να κάνει με τα ελαιούχα φυτά και την εθανόλη, βιοεθανόλη η οποία φτιάχνεται περισσότερο από ενοπνευματόδη. Προβλέψαμε λοιπόν ότι καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη την, ε, τις επιπτώσεις αυτών των καλλιεργειών στην έμεση αλλαγή της χρήσης γης. Αρχικά το Κοινοβούλιο Είχε μια προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμενόταν το 2010 να υποβάλει μια ε, έκθεση για το πώς ε, επηρεάζεται η χρήση της γης από τα στοιχεία αυτά και για το συντελεστή κάζι και κατά πόσον αυτό μπορεί να προσμετράται. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο κληθήκαμε να, να τοποθετηθούμε σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόταση η οποία Στόχο έχει να θέσει ένα ανώτατο όριο για τα βιοκάψιμα πρώτης γενιάς που προέρχονται από τέτοιες καλλιέργειες. Όμως, ο συντελεστής Κάζη θα υπολογίζεται μόνο στο επίπεδο υποβολής εκθέσεων και για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς τα οποία πρέπει να προωθηθούν θα υπάρξουν κίνητρα ώστε να φτάξουμε την ε, το 10%, 5% δηλαδή βιοκαύσιμα πρώτης γενναίας και 5% της δεύτερης γενναίας, χάρη ακριβώς ε, στη χρήση βιοκαυσίμων. Στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών ήδη είχαμε αρκετές ε, διαβουλεύσεις εντατικές και ξέρετε ότι και άλλες επιτροπές ασχολούνται με το κείμενο αυτό, με την πρόταση. Πολλά θέματα εφήγησαν. Πρώτα απ' όλα αυτό των ανώτατων ορίων και των στόχων που έχουμε θέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα ανώτατο όριο 5% για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενεάς. Παρόλο που δεν είχα ε, θεωρήσει καλύτερη αυτή τη λύση στην αρχική μου έκθεση, εγώ θα σας έλεγα να παραμένουμε στο 5% παρόλο που γνωρίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι θα θέλουν να ήμασταν περισσότερο φιλόδοξοι από το 5%. Όμως, συμπεριλαμβάνοντας το 5% αυτό τα βιοκάψιμα πρώτης γενεάς και τα μη εδόδημα φυτά για ενεργειακές χρήσεις, σημαίνει ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη τη χρήση γης σαν να επρόκειτο για καλλιέργεια εδόδημων φυτών. Θα έπρεπε να έχουμε έναν δευτερογενή όμω στόχο για τα βιοκάψιμα δεύτερης γενεάς με κάποιε λεπτομέρειε και διευκρινήσει σε σχέση με αυτό που πρότεινε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε διπλή ή τετραπλή προσμέτρηση ανάλογα με την κατηγορία βιοκαυσίμων. Κάποιες λίγες φορές διπλή και συνήθως τετραπλή προσμέτρηση. Εγώ προτείνω να έχουμε τη διπλή προσμέτρηση για όλα τα βιοκαύσιμα που αναφέρονται στο παράδειγμα 9 εκτός από τα φύκια και τα αερούχα ε, βιοκάσιμα βιολογικής προέλευσης, τα οποία θα χρησιμοποιούνται στις μεταφορές. Οι δύο αυτές κατηγορίες βιοκαυσίμων. Τέτραπλή προσμέτρηση για αυτά, διότι είναι τα πλέον προηγμένα. Χρειάζονται πολλές επενδύσεις για αυτά και ακριβώς είναι εκείνα που είναι πιο ελπιδοφόρα και διαταράσσουν λιγότερο άλλες, ε, άλλους κλάδους και τομείς που μπορούν να επηρεαστούν. Σας προτείνω όμως από το στόχο αυτό να αφήσουμε εκτός τα ζωικά λύπη διότι πρόκειται για προϊόντα τα οποία δεν ε, είναι θετική, δεν θετική ενθάρρυνση, βρίσκονται ήδη στην αγορά και τα έλεα ε, βιολογικής χρήσης έχουν ε, αποτελέσει και αντικείμενο απάτης. Πρόκειται για φυτικά έλαια, τα οποία συνήθως δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται καθόλου. Εδώ λοιπόν έχουμε το ανώτατο όριο και τους στόχους. Ε, σας είπα ποιες είναι οι λεπτομερείς, οι δευτερογενείς στόχοι. Τώρα υπάρχει ένας δευτερογενής στόχος ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Όπως έλεγα προηγουμένως, το 10% έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι μόνο τα βιοκαύσιμα λοιπόν. Γι' αυτό το λόγο προτείνω να υπάρξει ένας δευτεροτενής στόχος, δευτερογενής στόχος 1,5% για την ηλεκτρική ενέργεια προέλευση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται στα οδικά οχήματα και στους σιδηροδρόμους. Αυτό είναι συνεπές με το στόχο που έχουμε θέσει. Εάν προσθέσουμε το 5% βιοκαυσίμων πρώτης γενναίας και το 1,5% για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τρία για τα βιοκαύσιμα, τα προηγμένα που εξήγησα προηγουμένω, και το 1% των ζωικών λοιπόν και των οικοκυρικών ελαίων φυτικής προελευθή, θα έχουμε τελικά το 10%. Ένα συνεπή και ρεαλιστικό στόχο. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα. Κάζει. Αυτό θα πρέπει να το δούμε από δύο σκοπιές πιστεύω. Πρώτα απ' όλα από την άποψη της υποβολής εκθέσεων και έπειτα από τη συμπερίληψή του στα κριτήρια αηφορίας. Σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων προτείνω Όπω έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να το λάβουμε ευθύ αμέσω υπόψη. Γιατί, πρώτον, διότι ακόμη κι αν ορισμένοι συζητούν ακόμη το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό ο συντελεστή αυτό, υπάρχει ευρεία ε, συνένεση στο ότι υπάρχει ο συντελεστή αυτό. Είναι υπαρκτό. Εκεί που ξεκινά να συζητιέται το θέμα είναι πώ θα προσμετράτε. Το γεγονό όμω ότι έχει επίπτωση η χρήση της γης σε σχέση με την καλλιέργεια των φυτών βιοκαυσίμων και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στα αέρια του θερμοκηπίου, βεβαίως αυτό είναι αναντήρητο. Οπότε, πάνω απ' όλα για τους συναδέλφους που είναι πολύ προσεκτικοί στα επιστημονικά πορίσματα και θέλουν να είναι το θεμέλιο της ε, ε, νομοθετικής μας δράσης. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη και, για χάρη κοινων. Κατά δεύτερον, δεν πρόκειται για αλλαγή πολιτικής. Όπως προείπα, από το 2009 είχαμε ψηφίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι γνωστό και στο Συμβούλιο. Ε, έπειτα δεν είμαστε μόνοι στον πλανήτη και άλλες χώρες λαμβάνουν υπόψη το συντελεστή αυτό, ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά ή στα, στην Καλιφόρνια, στο, στην πολιτεία της Καλιφόρνιας ή η Βραζιλία. Και έπειτα για τις διαφορετικές τάσεις ως προς την προσμέτρηση, υπάρχει ένας τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε. Να ε, υπολογίσουμε και βάσει των ε, διαπιστωμένων αποτελεσμάτων, το συζητήσαμε με την κυρία Κλάση το πρωί και ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, να δούμε κατά πόσον αυτό που υπολογίσαμε είναι ορθό. Γι' αυτό το λόγο προτείνω άμεση εφαρμογή της ε, διαδικασίας υποβολής εκθέσεων. Το 2018 όμως να συμπεριληφθεί ο συντηλεστής ε, κάζε στο κριτήριο αηφορίας ώστε τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα στη βιομηχανία να προκύψουν ε, μετά το 2018. Δηλαδή αφού θα έχουμε ήδη στην διάθεσή μας μια τετραετία για να υπολογίσουμε ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις ε, από την συμπερίληψη του συντηλεστή κάζη. Κατά τρίτον, όπως όλοι, είμαι ιδιαίτερα προσεκτική με το τι συμβαίνει στην βιομηχανία και βεβαίως τις θέσει εργασία της βιομηχανίας της Ευρώπης. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσε επενδύσεις, ακόμη και αν πρέπει να παραδεχτούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων που γίνονται στον τομέα των βιοκαυσίμων έχουν καλυφθεί από του φορολογωμένου και όχι μόνο από τους ίδιους τους ε, φορεί τη βιομηχανία. Γι' αυτό σας προτείνω σας προτείνω να δούμε τι αντίκτυπο έχει ο συντελεστής Κάζη στις επιχειρήσεις έως το 2020 περίπου. Να θυμίσω και μόλις ακούσαμε τον κύριο Σίτερ, τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για το επιστημιστικά δικαιώματα να μας θυμίζει ότι οι πολιτικές που έχουμε χαράξει ως τώρα για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενεάς είχαν σοβαρότατο αντίκτυπο στην τιμή των τροφίμων και στην αρπαγή γεών σε περιοχές του Νότου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον μπορούμε να διατηρήσουμε μια τέτοια πολιτική και να δημιουργούμε μια βιομηχανική πολιτική που τη θέλουμε να είναι βιώσιμη, με... ενώ ταυτόχρονα προωθούμε προγράμματα όπως το Fit for Food. Για το βιοντίζελ λοιπόν προσφέρουμε πάνω από 50% των πρώτων υλών μας, ε, συμπεριλαμβανομένης της που χρησιμοποιείται στην Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο μου φαίνεται ε, λογικό να σας προτείνω να αναβάλουμε τον συντελεστή Κράζη κατά την συμπερίληψή του στο 2018 με μία περίοδο ε, ως το 2020 για το βιοντίζελ. Και θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τη μελέτη του συντελεστή Κράζη. Σε ό,τι αφορά την πορεία του FQ2. Σας προτείνω ένα 3% για το 2020 με το βιοντίζελ με ε, εθανόλη 6% το 2025, 9% το 2020 και 3% το 2018. Και αυτό για να μην ε, πληγούν τα κράτη που έχουν μεγαλύτερους στόχους για το 2018. Θα πρέπει να υπάρχει εδώ μια ρήτρα ευελιξία σε σχέση με το στόχο του 10% εφόσον τα κράτη αυτά ε, εκπληρώνουν τους στόχους ε, της Βασιλείας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές ήταν οι ανδρές γραμμές των συμβασμών που ήθελα να προτείνω. Γνωρίζω ότι τελικώς δεν είναι ακριβώς οι προτάσεις ούτε των μεν ούτε τον δε. Ελπίζω όμως ότι είναι ε, μια μεσαία, μέση λύση η οποία θα μας επιτρέψει να φτάσουμε με λογικές προτάσεις μας στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεπάς. Ήταν εκτενέστατη η εισαγωγή αυτή, αλλά όντως και το θέμα το ίδιο είναι πολύ ευρύ και ε, πολύ διαφορετικές αντιλήψεις και στο Κοινοβούλιο επ' αυτού. Ερχόμαστε τώρα στους κοιόδης συγητές από ε, τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Πρώτη εγώ, γιατί είμαι σκιώδη συγχύτρια του ΕΛΚ, την χάνω. Πολλές είναι οι τροπολογίες ε, που έχουμε. Ε, είναι ένα μπουκέτο πολύχρωμο αυτό μια ευρύτατη γκάμα και σκοπός είναι τώρα να συγκεράσουμε τις διάφορες απόψεις. Οι τόσο διαφορετικές ε, τροπολογίες δείχνουν ότι χρειάζεται ακόμα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και ευχαριστώ πολύ κυρία Λεπάς που δηλώνετε πρόθυμη και σήμερα και αύριο θα το συζητήσουμε αλλά και στη συνέχεια. Λοιπόν, χωρίς ε, περιστροφές θα έρθω στα βασικά σημεία που αναφέρατε κι εσείς. Πρώτον, ο υπολογισμός ε, ε, των διαφόρων παραγόντων σύμφωνα με το μοντέλο ΙΦΡΙ. Οι αλλαγές χρήσης γης ε, δεν είναι ε, θετική επιστήμη. Το έχουμε συζητήσει. Το φαινόμενο δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε άμεσα, ούτε να το μετρήσουμε άμεσα και ε, υπολογισμοί, μοντέλα και σε αυτή τη μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για τις επιστημιστικές πολιτικές δείχνουν ότι είναι πολλά τα κενά αλλά και τα σφάλματα ενδεχομένως στη μελέτη αυτή. Ε, άρα παραμένουν οι ασάφειες και βασίζονται σε κάποιες παραδοχές που είναι υποθετικές. Ε, θα πρέπει να το δούμε και από άλλη πλευρά και από άλλη σκοπιά το θέμα η μελέτη και το μοντέλο υπολογισμού ε, είναι και πάρα πολύ θεωρητικά και πάρα πολύ άσκηση επιχάρτου για μένα. Δεν είναι αυτό ε, πολιτική ε, με υπευθυνότητα. Και αν μας λέτε κύριε Λεπάζα, το αναβάλουμε μέχρι το 18, η μελέτη αυτή του ΙΦΠΡΙ παραμένει. Αλλά τη θεωρώ άγουροι, πώς να το πω, δεν είναι αρκετά όρημη για να μπορέσουμε να βασιστούμε και να αποφασίσουμε αργότερα. Ε, θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε αυτό και τον τρόπο υπολογισμού. Προσπάθησα στις δικές μου τροπολογίες να τα γράψω όλα αυτά και να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα υπολογισμού ε, που να βασίζονται στα πραγματικά στοιχεία αλλαγής γης και όχι σε υποθέσεις. Και επίσης για τα βιοκαύσιμα ε, σε αντίθεση με το μοντέλο του ΙΦΠΡΙ δεν βασιζόμαστε σε προγνώσεις, αλλά σε πραγματικά στοιχεία και ε, αλλαγές ε, χρήσης γης. Και αυτές οι τεχνικές δυνατότητες και οι στατιστική μας επιτρέπουν ε, ουσιαστική μελέτη. Τα άλλα στοιχεία μπορεί να είναι απαραίτητα, όπως ε, οι πρόταση ύλε, τα βιοκαύσιμα, η παγκόσμια γεωργική παραγωγή, όλα αυτά τα στοιχεία τα έχουμε και για τις καλλιέργειες και για το καύσιμο. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό που προτείνω εγώ στις δικές μου τροπολογίες, κάθε χρόνο βάσει πραγματικών στοιχείων γίνεται ένας νέος υπολογισμός. Το μοντέλο του ΙΦΠΡΙ ε, ορίζει ένα στατικό μοντέλο το οποίο δεν αλλάζει ούτε προσαρμόζεται από χρόνο σε χρόνο. Μα είναι μεταβλητές τα στοιχεία αυτά. Πώς θα κάνουμε αλλαγές αν είναι στατικά αυτά που δανειζόμαστε ως παραδοχές. Ε, θα πρέπει να κάνουμε σωστούς υπολογισμούς, να είμαστε υπέρ της βιωσιμότητας και να δημιουργούμε και κίνητρα. Γι' αυτό κάθε χρόνο χρειάζεται νέο υπολογισμός κατά την απόψή μου. Και κοινό μα στόχο είναι ακριβώ οι αλλαγέ χρήση να αποφεύγονται και κυρίω να μην αποψηλώνονται τα παρθένα δάση ε, ή να μην χάνονται υγρότοποι ε, ας πούμε και άλλοι πολύτιμοι ε, βιότοποι για την καλλιέργεια τέτοιων φυτών. Και πραγματικά αυτά θα πρέπει να μπουν ως βασικές πηγές. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν χώρες με άλλα πρότυπα και άλλα κριτήρια που δεν τηρούν ε, περιβαλλοντικά πρότυπα και να μην λέμε, να πούμε μάλλον ότι τα καύσιμά τους αυτά δεν είναι ευπρόσδεκτα στην Ευρώπη γιατί δεν τηρούν τους δικούς μας στόχους και πρότυπα. Πολλοί συνάδελφοι όπως και εγώ ζητούμε ένα ελάχιστο ε, στόχο 2% για τα προοδευτικά λεγόμενα βιοκαύσιμα. Ε, δηλαδή είναι και επενδυτικό κίνητρο αυτό και πιο σκόπιμο από ένα τέτραπλό ή διπλό ε, υπολογισμό ή προσμέτρηση. Αυτό οδηγεί και σε στρεβλώσεις της αγοράς και αλλάζει και το στόχο, ξεφεύγει από το 10% το ε, ανανεώσιμο στις μεταφορές. Μα εμείς πώς θέλουμε να φτάσουμε στους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον και στις μεταφορές. Αν είναι δεσμευτικοί οι στόχοι για τη δεύτερη πλέον γενεά, Δημιουργούνται έτσι προϋποθέσεις και κίνητρα για να παράγονται αυτά τα καύσιμα και πρέπει να προσαρμόζεται και η τεχνολογία γιατί δεν είναι όλα πια τόσο ε, όριμα και εξελιγμένα. Νομίζω θέλει προσοχή εδώ. Όταν έχουμε τετραπλούς ε, υπολογισμούς είναι δεύτερη γενεά, δεν είναι από πρώτο χέρι, είναι μεταχειρισμένο με το εμπόρευμα και μπορούμε να το παράγουμε. Ε, χρησιμοποιούνται, μου είπαν πολλοί όλα αυτά ε, ουσίες, δεν είναι υποπροϊόντα, είναι παραπροϊόντα, δεν είναι απόβλητα δηλαδή, τα χρησιμοποιούμε. Και σε κάθε οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, στόχος μας είναι ο περισμός των αποβλήτων ε, έτσι, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ε, χρειαζόμαστε ένα συνδυασμό μεταξύ αυτών των τριών στοιχείων. Εκεί είναι το κλειδί. Δηλαδή, ο πρώτος, ο στόχος ε, οροφής, ε, ε, η νέα διαδικασία υπολογισμού του ανωτάτου ορίου για τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από καλλιέργειες για να αποτραπεί αλλαγή χρήση γης, αλλά να ξεκαθαρίσουμε και γι' αυτό είναι σημαντικό για μένα ότι και η ευρωπαϊκή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μεταφορές δεν θα πρέπει να καταστραφεί. πρέπει να παράγουμε και εμείς τη δική μας ενέργεια, να μην εξαρτώμαστε πάντα από τρίτες χώρες. Έτσι αυξάνεται και η ε, ανεξαρτησία μας από αμφίβολες και επισφαλείς ε, προμήθειες ε, από τρίτες χώρες. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κάνει και τροπολογίες και φαντάζομαι ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό κοινό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ και θέλω να δώσω το λόγο τώρα στους υπολείπους σκιώδης ηγητές. Ο κύριος Αρσένης από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, παρακαλώ. Thank you very Σας κατευχαριστώ. Νομίζω ότι η θέση μας πρέπει να βασίζεται σε τρεις αρχές. Η μία είναι να μην χρησιμοποιούνται δημόσιες επιχορηγήσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών για προγράμματα και προϊόντα που δεν οδηγούν σε εξοικονομήσεις αλλά χρησιμοποιούν περισσότερες εκπομπές που βλάπτουν το περιβάλλον. Αυτή είναι μία βασική αρχή. Δεύτερη αρχή. Να αντιμετωπίσουμε μία τρομακτική επίπτωση αυτών των προγραμμάτων και πολιτικών που δημιούργησε μεγάλη ανέχεια σε πολλά μέρη του κόσμου όπου η κατάσταση είναι ήδη δύσκολη. Και τρίτον, να προστατευθούν οι υπάρχουσες επενδύσεις. For the Για να διαχωρίσουμε μεταξύ καλών και κακών βιοκαυσίμων πρέπει να φανεί ότι τα 10 δισεκατομμύρια ετησίων επιχορηγήσεων άμεσων και έμεσων προς τα βιοκαύσιμα, προς τη βιομηχανία των βιοκαυσίμων, δεν οδηγούν σε περισσότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αυτό πρέπει να δείξουμε. Ότι δηλαδή το, η πραγματική επίπτωση της παραγωγής κάθε είδους βιοκαυσίμου να δείχνει αν ωφελεί ή όχι και να φαίνεται ότι οι δημόσιες επιχορηγήσεις οδηγούν σε εξοικονομήσεις ε, εκπομπών, όχι περισσότερες. Για τα αγροτικά τώρα, για τις Ο κύριος Δεσούτα και η κυρία Λαπάς ναι. είπαν ότι ο εκπρόσωπος της ΦΑΟ μας μίλησε πριν από μερικές εβδομάδες και είπε ότι οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, τα όργανα του ΟΗΕ, επανειλημμένως δήλωσαν ότι η πολιτική αυτή της Ένωσης οδήγησε άμεσα σε αύξηση των παγκοσμίων τιμών ή των τιμών παγκοσμίω. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη γεωργία έτσι. Τι πείνα. Γιατί έτσι δημιουργείται ανέχεια και πείνα. Όπως είπε και ο κύριος Σούτε και όλοι οι άλλοι, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις επενδύσεις, γιατί υπάρχουν επενδύσεις για τα βιοκαύσιμα, χρησιμοποιούν το 4,8% των καλλιεργιών. Το ανώτατο όριο του 5% λοιπόν βοηθάει στην καταπολέμηση των εκπομπών και προστατεύει τις επενδύσεις. Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι είχα προτείνει τον πολλαπλασιαστή 2,5 για τα ηλεκτρικά τρένα. Η πρόταση της κυρίας Λαπάζ είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα τη συζητήσουμε όπως πρέπει. Τέλος, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε βιοκαύσιμο δεύτερης γενεάς πρέπει να παράγεται μόνο με περισσεύματα. Αυτό πρέπει να είναι σαφές για όλη την παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς. χωρίς τρύπες στην νομοθεσία. Αλλιώς θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Πρέπει να αποσαφινιστεί ότι θα χρησιμοποιούνται τα περισσεύματα γενικά. Um, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ την εισηγήτρια Κορίν Λεπάζ για την θέση της για τα βιοκαύσιμα που είναι λεπτό θέμα γιατί 7 επιτροπές γράφουν γνωμοδοτήσεις και έκθεσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Δεν θα είναι εύκολο. Αύριο η Ήτρε θα ψηφίσει. Και αν δει κανεί προς τα που κινείται καταλαβαίνει γιατί ανησυχώ διότι οι συνάδελφοι που ακούν επιστήμονες ή όπως είπε και ο Κρήτον, ο, τον Ολιβιέντε Σότερ, συμφωνούν ότι υπάρχει πρόβλημα, κάτι πρέπει να αλλάξει, όχι όμως τώρα. Και συνεχίζουν τα πράγματα χωρίς καμιά αλλαγή. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν έλλειψη αξιοπιστίας για το Κοινοβούλιο αν δεν κάνουμε κάτι για τα βιακάψιμα. Γι' αυτό σας υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από την Επιτροπή να κάνει κάτι. Στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο είχαμε υποχωρήσει βέβαια και γι' αυτό καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική διατύπωση όπου έλεγε παρακαλούμε την Επιτροπή να κάνει μια ανάλυση και μια πρόταση. Η Κομισιόν το έπραξε. Έκανε την εκθέση της και πρότεινε κάτι. Αλλά και στην Επιτροπή υπήρξαν παρόμοιες διαμάχες όπως το Κοινοβούλιο και γι' αυτό κατέληξαν σε μία ασαφή πρόταση. Να υπάρξει ένα όριο στη βιοκάψιμα πρώτης γενεάς και να μην κάνει τίποτα συγκεκριμένο και άμεσα. Κάτι πολύ ασαφές δηλαδή, γιατί αν συμφωνούμε όλοι ότι η αέμεση χρήση της γης είναι πρόβλημα και τώρα μας λένε ότι δεν είναι πρόβλημα ή ότι πρέπει να κάνουμε κάτι αλλά δεν γνωρίζουμε ότι η αδράνεια θα σημαίνει παράγοντα μηδέν Αυτό ετοιμάζουμε τώρα uh, για το ILOC. Όσοι λένε ότι αλλάζουν έτσι όλοι οι κανόνες, θα ήθελα να σας πω ότι στη συζήτηση αυτή, η συζήτηση αυτή υπάρχει εδώ και 5-6 χρόνια. Και επομένως οι επενδυτές ήξεραν ότι θα γινόταν αυτή η συζήτηση, ότι υπάρχουν προβλήματα με την πρώτη γενεά βιοκαυσίμων και ότι ήταν πολύ πιθανό να αντιδράσει η Ένωση. Αυτά γενικά, αλλά το θέμα είναι τι θα αποφασίσουμε. Το κυριότερο είναι τι θα κάνουμε τα τωρινά βιοκαύσιμα πρώτης γενεάς. Η Κομισιόν προτείνει λοιπόν όριο 5%. Ξέρω ότι αύριο στην Ήτρε θα γίνει μια συμβιβαστική πρόταση 6,5% το οποίο είναι σχεδόν business as usual και η πρόταση τώρα στην περίφ είναι να διατηρηθεί αυτή η πρόταση του 5%. Αλλά τι κρύβουν όλα αυτά. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται από καλλιέργειες και τα άλλα. On less productive lands. But if you are... Μερικά φυσικά θα συνεχίσουν να βασίζονται στις καλλιέργειες, αλλά αν θέλουμε πιο παραγωγικές γέες ή όχι, τι θα διαλέξουμε ακόμη και για το βουτρόφα. Ε, φυτό είναι και αυτό. Χρειάζεται γη. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε τα βιοκαύσιμα από καλλιέργεια και μη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει η χρησιμοποίηση των βιοκαυσίμων και από τις καλλιέργειες των φυτών καθε αυτά. Υπάρχουν λοιπόν από την άλλη μεριά και τα βιοκαύσιμα που δεν προέρχονται από χρήση γης. Μόνο έτσι θα δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί για τα βιοκαύσιμα. Αλλά επαναλαμβάνω εννοώ βιοκαύσιμα που δεν βασίζονται στις καλλιέργειες είτε το γιουτρόφα είτε άλλων φυτών. Άλλη σημαντική συζήτηση που θα προκύψει είναι τι να γίνει μετά το 2020. Η Κομισιόν δεν μας έχει πει τίποτα γι' αυτό. Στην Ήτρε βλέπω ότι παρατείνουν τη διορία και μετά το 2020. Η Κορίν Λεπάζ είχε τη σοφία να προτείνει όντως μία διορία πέραν του 2020 γιατί το θέμα τίθεται. Θέλουμε την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, τη μείωση του διοξιδίου δηλαδή και τα ανανεώσιμα να τα συνδέσουμε με διορία 2020. Το πρώτο είναι τεχνολογικό στόχος, το δεύτερο τονίζει περισσότερο το στόχο της μείωσης του διοξιδίου. Ο τεχνολογικός στόχος δεν είναι ευέλικτος. Χρειάζεται να παραχθεί ο αλφα όγκος. Ό,τι και να συμβαίνει κρίση είναι η κρίση. Είναι μη ελαστικό στόχος λοιπόν. Γι' αυτό είμαι υπέρ μετά το 2020 να συνεχίσει η εφαρμογή της οδηγίας της ποιότητας των καυσίμων και όχι τόσο πολύ των ανανεωσίμων. Τέλος, για το ΆΙΛΟΚ. Τώρα έχει φανεί ότι πρέπει να αρχίσουμε να το παίρνουμε υπόψη μας, γιατί αν περιμένουμε άλλα πέντε χρόνια, οι ίδιοι επενδυτές θα μας πούν τώρα είναι όλα καινούργια και κάναμε λάθος επενδύσεις. Αυτοί θα συνεχίσουν να υπάρχουν όμως πάντοτε και δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αποσιάζουν οι συντηρητικοί και οι ευτοί, οπότε το λόγο έχει τώρα η Σαμπίνε Βίλς από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Λεπάζ. Οι συζητήσεις για τις δύο οδηγίες είναι μεγάλη πρόκληση γιατί θέλουμε καινοτόμε λύσεις με υφιστάμενους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παραγωγή των βιοκαυσίμων που μέχρι τώρα δεν είναι ε, πάρα πολύ βιώσιμη και αηφόρο. Η οδηγία ILOC ε, αμφισβητείται εν μέρη γιατί προσάπτουν στη μέθοδο να μην είναι ε, η σωστή ή να μην είναι για να φτάσουμε στους στόχους. Για τη δική μου πολιτική ομάδα έχει σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για να διατηρήσουμε τη γη μας, ε, για να καλλιεργούμε ε, ε, φυτά τα οποία προ ορίζονται για την παραγωγή τροφίμων και πολύ συχνά από μικρούς αγρότες. Ε, αποτελεσματικότητα θέλουμε και στην ενέργεια και χρειάζεται ανώτατο όριο για την παραγωγή παραδοσιακών βιοκαυσίμων και ένα στόχος για ε, τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς. στην Επιτροπή Μεταφορών που έχω κάνει τη γνωμοδότηση, ε, έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και προσπάθησα να θέσω τον ίδιο στόχο Υπήρξε μια επίμαχη συζήτηση εκεί για τα ανώτατα όρια μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων και για να συμφωνήσουμε ο συμβιβασμός λέει 6,5% και 3% για τη δεύτερη γενιά. Αυτό ζητάει η Επιτροπή Μεταφορών. Η δική μου πολιτική ομάδα συμφωνεί απολύτως όμως και με το συμβιβασμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τον υπολογισμό στο άρθρο 7 δέλτα θα πρέπει να ισχύουν ε, πάντα οι παράμετροι ILOC ε, και αν έχουμε νέα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2016 ε, τότε θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε καλύτερα. Να μην υπάρχει το λεγόμενο grandfather right μέχρι το 2025. Εγκρίθηκε λοιπόν αυτή η πρόταση και στην Επιτροπή Μεταφορών και στον μαθηματικό τύπο ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η τεχνολογία για την αξικονόμηση ενέργειας και για τη χρήση ε, ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Και το θέμα των αποβλήτων και των υπολοιμάτων είναι για μας πολύ σημαντικό. Τα βιοκαύσιμα που αναφέρονται στην παραγωγή δεν θα πρέπει να παράγονται από απόβλητα και υπολείμματα βάσει της οδηγίας του 2008 98 ε, ε, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Επίσης να βελτιωθούν οι συμφωνίες ε, με αυτόχθονες πληθυσμούς και κοινότητες για να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και τα δικαιώματά τους να προασπίζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει εκθέσεις ε, για, να αποφεύγει, για την παρακολούθηση όλων αυτών για να αποφεύγεται η αρπαγή γης, το λεγόμενο land grabbing και ελπίζω να καταλήξουμε όλοι οι σκιώδεις ηγητές σε ένα καλό αποτέλεσμα με ένα υφόρο κείμενο όσο και φιλόδοξο που θα καταθέσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ κυρία Βίλτς. Ολοκληρώνεται εδώ ο γύρος των σχεδόν εισηγητών και θα δώσω το λόγο. Θα καλωσορίζω και τον Αλέχο Βιδάλ Κουάδρας που έχει κάνει την έκθεση στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Να του δώσουμε το λόγο να μας πει τη γνώμη του κι αυτός. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι και πάλι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να σας αναφέρω τις εξελίξεις στη δουλειά μας, την Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας, για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ ξανά την Κορίν Λεπάζ για την καλή συνεργασία που είχαμε και τη γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Όπως τα γνωρίζετε, στην Επιτροπή Βιομηχανίας θα ψηφίσουμε αύριο. Και έχουμε αφοσιώσει πολλές προσπάθειες στην εξέδεση συμφωνίας που να μπορεί να στηριχθεί από την πλειοψηφία των μελών. Είχαμε επανειλημμένα συναντήσεις των σκιωδών 8-10 ώρες συζητήσεις κάθε φορά και στο τέλος καταλήξαμε σε μια συμφωνία για τα κέρια σημεία. Ελπίζουμε να τύχουν αρκετή στήριξη οι συμβασμοί μας αύριο. Ως προς τον συντελεστή ILOC. Η πλειοψηφία, όχι όλοι, η πλειοψηφία συμφωνήσαμε ότι δεν θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των εκπομπών. Συνεπώς, δεν θα υπάρξει υποχρέωση στο επίπεδο της υποβολής εκθέσεων. Όμως θα συστήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να υποβάλει εκθέσεις και να συγκεντρώνει στοιχεία και στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων που αυτή τη στιγμή είναι αρκετά αβέβαιες και αρκετά ασαφείς. Στο μέλλον λοιπόν να καταλήξει όλη αυτή η προσπάθεια σε μια συγκεκριμένη πρόταση για υποχρέωση στην υποβολή εκθέσεων. Ω προ το ανώτατο όριο για τα συμβατικά βιοκαύσιμα, είχαμε προτάσει 3-4% κάτω του 5% δηλαδή και δύο προτάσει για κανένα ανώτατο όριο. Στο τέλο η πλειοψηφία συσπηρώθηκε γύρω από το ανώτατο όριο του 6,5%. Ως προς τα προηγμένα βιογράψιμα, προτείναμε να θέσουμε ένα συγκεκριμένο δευτερογενή στόχο 2,5% για το 2020. Ως προς την πολλαπλή προσμέτρηση Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα να μην ληφθεί υπόψη, διότι θα θέσει ένα αμφιβόλο το συνολικό στόχο του 10%. Είναι σαν να κοροϊδεύουμε τους αυτούς μας, κάτι που θα είναι αντιπαραγωγικό μάλλον. Τέλον, τέλος, ε, προτείναμε μέτρα για την καλλιέργεια και την προώθηση της εθανόλης με ένα 5% κατανάλωσης πετρελαίου στο 2020. Ένα πολύ φιλόδοξο ενεργειακό μείγμα. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας μας. Συμφωνίας που όπως σας είπα προς βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι των σχεδόν εισηγητών. Η Επιτροπή έχει πολύ περισσότερα μέλη από ότι ο στενός κύκλος των σχεδόν εισηγητών. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αύριο στην ψηφοφορία. Πάντως καταρχήν έχουμε σοβαρές ελπίδες ότι θα υπάρξει πλειοψηφία αύριο και θα στηρίξει αυτές τις προτάσεις που μόλις σας παρουσίασα. Καταβάλαμε πραγματικά μεγάλες προσπάθειες για να συμβάσουμε τις διαφορετικές θέσεις μεταξύ τους. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι στην αρχή οι θέσεις ήταν, ε, απήχαν πόρο ημένα από του ΙΣΔΕ. Η προσπάθειά μας λοιπόν να βρεθεί τελικά μια συμφωνία ήταν εντονότατη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Αλέχο. Βιδαλκό Καλή επιτυχία για αύριο στην Επιτροπή σας αλλά και για την ουσία για το θέμα. Ωραία, οι υπόλοιποι, τέσσερις, ο Γιολάινα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κορίν Λεπάζ έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά για την έκθεση αυτή και όταν πιάνει ένα θέμα είναι πάρα πολύ μεθοδική και το δουλεύει σε πολύ μεγάλο βάθος. Και αυτό το θέμα, ε, το χρειάζεται αυτό γιατί είναι περίπλοκο. Ε, παράλληλα με εμά ταυτόχρονα στην άλλη πλευρά ε, του κτηρίου συνεδριάζει ισομερή συνέλευση ΑΚΕ και είμαι και εκεί μέλος κι εγώ και πρέπει να σας πω ότι από την Αφρική κυρίως μας παρακολουθούν πάρα πολύ στενά και από κοντά τι κάνουμε με τα βιοκαύσιμα γιατί οι τιμές των τροφίμων και η έλλειψη της γης είναι ένα θέμα που αφορά και την Αφρική αλλά και τις άλλες επίρους Από πλευρά στόχων θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν έχει νόημα να υποστηρίζουμε κάποιες δραστηριότητες και με χρήματα των φορολογουμένων μάλιστα που έχουν αρνητικές επιπτώσεις τελικά στο περιβάλλον και στην προστασία του κλίματος. Δεν επιτρέπεται να δίνουμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες επιβαρύνουν την κατάσταση και μας εμποδίζουν να φτάσουμε και στην καταπολέμηση και στην πάυση της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, αυτό το θέμα το ILOC είναι απολύτως απαραίτητο. Ε, κάτι άλλο που θεωρώ είναι ότι μας είχε πιάσει υπερβολική εφορία τότε όταν βάλαμε τόσο ψηλούς στόχους και ανώτατα όρια. Ε, γι' αυτό χρειάζεται τώρα οπωσδήποτε μια οροφή, διότι πρέπει λίγο να το συμμαζέψουμε και να το περιορίσουμε προς τα κάτω, ε, προς τα πάνω. Έχω όμως μια ανησυχία, γι' αυτό ζήτησα και το λόγο. Να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Δεν επιτρέπεται κατά την άποψή μου. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια συνεδριάζει ε, πανευρωπαϊκά μια οργάνωση αγροτών που ε, παράγουν βιοκαύσιμα προς ίδια χρήση οι αγρότες. Και στη διάσκεψη του Ντέρμπαν του ΟΗΕ είχα την ευκαιρία ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας να κάνω ένα site event εκεί και ε, είχε έρθει ο Τζον Τίρι, ξέρετε, η μεγάλη εταιρεία τρακτέρ. Είχαν βάλει ολόκληρο ε, ελκυστήρα, ε, το οποίο ο τρακτέρ έχει ως κάψιμο ένα σπορέλαιο. Λοιπόν, υπάρχουν αγρότες που καλλιεργούν αυτά τα φυτά και χρησιμοποιούν στα τρακτέρ τα κάψιμα από τα φυτά τους. Λοιπόν, δεν θέλω αυτή την προσπάθεια να την καταστρέψουμε με αυτά που θα προτείνουμε. Αξίζει να την υποστηρίξουμε υπάρχουν ε, παραγωγές μικρής κλίμακας δεν έχουν καμία τεράστια επίστοση στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως τώρα. Οι διαγρότες το κάνουν έτσι συμπροματικά. Παράγουν τρόφιμα και παράγουν και αυτά για να έχουν τα καύσιμά τους. Έχω κάνει και αντίστοιχες τροπολογίες ε, και θα πρέπει να φροντίσουμε και να καταλάβουμε ότι ορισμένα ελαιούχα φυτά είναι και πρωτεϊνούχα για τα ζώα ας πούμε ε, ε, είναι ένας πλακούντας τον οποίο χρησιμοποιούν στη συνέχεια για να ταΐζουν τα ζώα. Και μετά ε, το λάδι που παίρνουν όταν το χρησιμοποιούν για καύσιμο είναι καλό. Λοιπόν, να μην καούν και τα χλωρά μαζί με τα ξηρά και είναι μια ωραία βιομηχανία, ένας ωραίος κλάδος που γεννήθηκε τα τελευταία χρόνια και δεν θα πρέπει να το καταστρέψουμε αυτό με τα καύσιμα από ελαιούχα φυτά. Ε, ο πολλαπλός ε, υπολογισμός είναι ένα πρόβλημα γιατί το άκουσα κι εγώ. Για τελικά θα καταντήσουν τα αποβλήματα να είναι πιο ακριβά από ε, τον ίδιο το καρπό. Δηλαδή το άχυρο θα είναι πιο ακριβό από ότι το σιτάρι και έχω δει και κόσμο να ψάχνει άρον-άρον να συλλέγει άχυρα ε, για να έχει ε, αυτό το πολλαπλασιαστή και το αποτέλεσμα και να πάρει και πολλά λεφτά. Λοιπόν, ε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο τι κάνουμε για να μην δίνουμε λάθος κίνητρα και έχουμε στρεβλές καταστάσεις που μπορεί να ακούγονται ωραία. Τα βιοκαύσιμα λέει δεύτερης γενεάς, θαυμάσιο, αλλά όταν παράγονται τέχνητά τότε υπάρχει πρόβλημα και ανεπιθύμητες συνέπειες. Εκατοντάδες είναι οι τροπολογίες και ελπίζω οι σκιώδεις συζητητές να μπορέσουν να συμφωνήσουν για ε, λογικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε κύριος Παρνιό. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της πάνω σε αυτό το ιδιαίτερα πολύπλοκο και τεχνικό θέμα, όπως και πολιτικό. Δεν μπορούμε πια να επιλέξουμε μεταξύ οδήγησης και διατροφής. Και γι' αυτόν τον λόγο μεταξύ άλλων η συμπερίληψη του Καζή από την, του συντελεστή Καζή από την Κομισιόν ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Εχθές εγκρίναμε εμεί τη γνωμοδότησή μας και για να ενισχυθούν οι επενδύσεις και η απασχόληση θέσαμε το όριο της χρήσης των βιοκαυσίμων εκεί που το θέσαμε. Αυτές είναι και οι τροπολογίες, αυτά αφορούν και οι τροπολογίες που κατέθεσα. Η Επιτροπή Μεταφορών κατέληξε σε ορισμένες συμβιβαστικές που εγκρίθηκαν σχεδόν από όλες τις ομάδες και διασφαλίσαμε και τη συνέχιση της χρήσης των ε, βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς κατά 6,5% σε ποσοστό 6,5%. Να το πάρετε παρακαλώ υπόψη σας και εσείς. Πέρα από αυτό το όριο η Επιτροπή Μεταφορών προτείνει έναν στόχο υποστόχο 3% για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς ώστε μέχρι το 2020 να έχουν αναπτυχθεί. Μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε το παράδοξο η αγροτική κατανάλωση να βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την κατανάλωση για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Αύξηση των τιμών, αποδάσωση ήταν οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να εγκρίνουν ένα κείμενο που νομίζω ότι αντιμετωπίζει σωστά το πρόβλημα και με υπευθυνότητα και προς τις επιχειρήσεις κυρία Πρόεδρε μου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκροστέτ, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Δεδομένου ότι πολλά έχουν ήδη καλυφθεί, θα επιμείνω σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα στην έκθεση της η κυρία Λεπάζ να προβλέψει την ενθάρρυνση της ερεύνας για τα βιοκαύσιμα. Να θυμίσω εδώ ότι το μεγαλύτερο μέρος του στόλου των ε, οχημάτων στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το βιοντίζελ. Άρα σε πρώτη φάση σημαντικό είναι να έχουμε σημαντικές ποσότητες βιοντίζελ, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε και την ε, χρήση που είναι, ήδη γίνεται στα αυτοκίνητα. Μην δυσκολέψουμε τους συμπολίτε μας. Δεύτερη παρατήρηση θα ήθελα να ληφθεί περισσότερο υπόψη τι πηγές χρησιμοποιούμε και μάλιστα πηγές που δεν ανταγωνίζονται την παραγωγή τροφίμων, όπως τα φύκια ή τα ξυλοκυταρικά κατάλοιπα δασοκομικής προέλευσης, τα οποία σήμερα δεν αξιοποιούνται επαρκώς είναι ε, σημαντικότατες πηγές αυτές σε πολλά κράτη-μέλη. Ε, έχουμε πολλά σημαντικά κοιτάσματα και σε συνεργασία με πολλούς Γαλλούς συναδέλφους υπέβαλα σχετικές τροπολογίες. Βρίσκεται βέβαια σε πρωτογενές στάδιο η όλη προσπάθεια και η χρήση της πηγής αυτής, όμως έχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η σχετική έρευνα. Θα ζητούσα από την κυρία Λεπάς, της οποίας χαιρετίζω φυσικά τη δουλειά, να πει κάτι και για αυτά τα βιοκαύσιμα δεύτερη γενναίας με τη χρήση μεταξύ άλλων των καταλήπων βιομάζας και αυτέ ήταν οι παρατηρήσει τι οποίε ήθελα να σα επισημάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μασέη Κούκοβιτ, και μετά ο Κασούτα τελευταίο. Uh, thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές, διότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Από πολλές διαφορετικές σκοπιές. Κατά πρώτον, να πω ότι χρειάζεται περισσότερη ανεξαρτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για τις διαφορετικές πηγές ενέργειας, αυτό πρέπει να το έχουμε διαρκώς κατά νου. Ταυτόχρονα ωστόσο, όταν μιλάμε για βιοκάψιμα που σχετιζόνται με τη χρήση γης, δεν μπορούμε τώρα να αποκλείσουμε αυτού του είδους τα βιοκάψιμα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα οι γεωργοί, οι οποίοι ζουν στις καλλιεργόμενες περιοχές. Δεν μπορούν να αλλάζουν ε, μια ανοιχτή τις στρατηγικές τους, τις στρατηγικές καλλιέργειες πρέπει να χρησιμοποιήσουν απλώς τις γόνιμες γεές που είναι καλλιέργητες. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία σε πολλά κατημέλη, ιδίως στη Σλοβενία. Υπάρχουν λοιπόν ε, χιλιάδες επί χιλιάδων ε, εκτάρια τα οποία είναι ακαλλιέργητα και χρησιμοποιείται. Αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους γεωργούς αλλά και για την ε, βιομηχανία, το σχετικό κλάδο. Σήμερα έχουν στα χέρια τους τις καλύτερες, τα καλύτερα δυνατά τεχνολογικά μέσα, αλλά δεν υπάρχουν χώροι εργασίας. Ταυτόχρονα έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία δεν έχουν σταθεροποιηθεί και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ακόμη ως ε, ενεργειακή πηγή. Η λάσπη λοιπόν από απόβλητα, η λιματολάσπη, θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να διασυνδέσουμε την βιομηχανία με τις ενεργειακές πηγές, να τους διευκολύνουμε. Εδώ προσφέρονται πολλές ευκαιρίες, ίσως κάποιες διαφο κάπως διαφορετικές από αυτές που σήμερα βλέπουμε, αλλά πρέπει να έχουμε και πολλές διαφορετικές απόψεις για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη γη χαρακτηρισμένη ή όχι. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές πηγές για όλους μας. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ακόμη υπάρχει τεράστια εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα στην Γεωργία. Και να σκεφτούμε ποια εδάφη θα χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια τροφίμων, εφόσον δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πλέον ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή λιπασμάτων. Ποιοι αγρότοποι θα χρησιμοποιούνται για τα καύσιμα και ποιοι για τα τρόφιμα. Το ίδιο και τα δάση. Νομίζω η εισηγήτρια έχει προσεγγίσει πολύ καλά το θέμα και έχει εξηγήσει με ε, εύστοχο τρόπο το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται και τα ε, δάση, αλλά τα ίδια τα δέντρα και καρπίτους τους, όπως η συλλογή και η συγκομιδή μούρων και βατόμουρων. Είναι σημαντικό αυτό από τη σκοπιά της χρήσης ενός δάσους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό του είδους τις αξίες που είναι πιο παραδοσιακές. Επιπλέον, εγώ ίδιο στην πανεπιστημιακή μου σταδιοδρομία ασχολήθηκα με το θέμα των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα με τη χρήση τεχνολογικών μέσων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Εάν λοιπόν παίρναμε απόβλητα όπως η λιματολάσπη και μπορούσαμε από αυτή να παράγουμε αέριο, σίγουρα θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ενεργειακή περιεκτικότητα των καυσίμων αυτών καθεαυτών. Ούτε θα χρειαζόταν τόση μεταφορά λιματολάσπη. Διπλό το κέρδο λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θα κερδίζαμε ενέργεια και μετά θα τη χρησιμοποιούσαμε με φτηνότερο κόστο. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε κατά νου αυτό. Πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα απόβλητα. Δεν μπορούμε όμω να τα θέλουμε όλα ταυτόχρονα και να τα πετύχουμε και ταυτόχρονα για τα βιοκάψιμα πρέπει να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους και να δούμε πώς θα επηρεαστεί η χρήση της γης, εάν θέλουμε περισσότερα βιοκάψιμα. Άρα, νομίζω, εδώ υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των, αποβλη... των αποβλήτων, ώστε με ένα σπάρο να έχουμε δύο τριγώνια. Η εισαγήτρια πάντως έχει πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε με τρόπο άριστο και στο μέλλον για το στόχο μας. Ευχαριστώ. Κυρία Μέρκη ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, τα βιοκαύσιμα μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία ε, απέναντι στην εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, αλλά θα πρέπει να δείξουμε προσοχή και να είναι ευκαιρία και όχι τμήμα του προβλήματος από ό,τι φάνηκε τελευταία. Ε, και συμφωνώ με ε, την οροφή που προτείνεται, το 5% και το ILOC, ε, ε, αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι 800 εκατομμύρια τόνους διοξίδιο του άνθρακα ε, η οροφή που είναι ποσό που αντιστοιχεί στις εκπομπές της Γερμανίας. Όταν έχουμε 10% ανανεώσιμες μόνο με διπλό υπολογισμό Νομίζω δεν είναι σωστό. Καλό είναι να έχουμε ένα ουσιαστικό γνήσιο υποστόχο. Εγώ προτείνω ένα 3%. Και επίσης τα βιοκαύσιμα δεν είναι μόνο τα μόνα βιώσιμα καύσιμα ή φαίνεται να είναι. Ε, έχω προτείνει να κοιτάξουμε και άλλα καύσιμα μεταξύ αυτών. τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα, ας πούμε, βέβαια να έχουν παραχθεί με βιώσιμες πηγές ε, ε, κάθε φορά ε, ε, η ενέργεια, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα. Πριν από 10 χρόνια θεωρούσε κάποιος ότι τα βιοκαύσιμα είχαν μόνο πλεονεκτήματα για ανθρώπους στην Αιθιοπία, την Ταζανία κτλ. Και τώρα βλέπουμε τεράστια προβλήματα. Τους αρπάζουν τη γη και καταπατούν τα δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων. Αυτά θα τα δούμε και στην έκθεση, έχω κάνει τροπολογίες και θέλω πραγματικά να υπάρχει αηφορία αλλά και μέρημνα κοινωνική. Η κυρία Σοφία Κονή ζήτησε τώρα το λόγο, αλλά κλείνω τον κατάλογο και μετά θα μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη Σοφία Κονή. Δεν θα επαναλάβω όσα υπόθηκαν. Συμφωνώ με πολλούς από τους συναδέλφους και ήθελα πραγματικά να χαιρετήσω το έργο της κυρίας Λεπάζου. παρόλο που δεν έχω μελετήσει κατά λεπτό το όλο θέμα, καταλαβαίνω πόσο σοβαρά και περίπλοκα είναι τα θέματα που μελέτησε. Για το 10% λοιπόν του αρχικού στόχου. Αγαπητή Κορίνα, αναρωτιέμαι, με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε, θα μπορέσουμε να επιδείχουμε αυτό το στόχο τελικά. Ξέρουμε ήδη κάποιοι μπορούμε από τώρα να το φανταστούμε. Ο στόχος αυτός θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Και αυτό είναι και το αντικείμενο της τροπολογίας που υπέβαλα. Καλό θα ήταν επιτέλους να έχουμε στόχους που να μπορούμε να επιτύχουμε και να μην είμαστε υποκριτές ως προς τον εαυτό μας, να προτείνουμε πράγματα που δεν είναι εφικτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη παρατήρηση δεν έχει να κάνει ακριβώς με τα βιοκαύσιμα αυτά καθεαυτά, αλλά με την προβληματισμό που πρέπει να αναπτύξουμε και να αποφασίσουμε αν θα οδηγούμε ή θα έχουμε τρόφιμα έκθεση που δημοσιεύτηκε εδώ στο Κοινοβούλιο από τον κύριο Ντοντά, τον συνάδελφο, για την ε, ε, επιστηστική σπατάλη, τη διασπάθηση των επιστηστικών πόρων. Στην ε, παραγωγή λοιπόν τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 50% της παραγωγής δεν αξιοποιείται. Έχουμε τόσο σοβαρά ζητήματα και τόσο σοβαρά ντοσχεία όπως αυτό. Δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικέ λύσεις για τα ορυκτά καύσιμα, σίγουρα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μελετήσουμε και να επιδιώξουμε την εφαρμογή των κειμένων όπως αυτού που δημοσιεύτηκε και αυτά όχι μόνο να διακοσμούν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τα γραφεία των Υπουργείων κάποιων κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη η ψαλίδα και το φάσμα ε, των απόψεων και με πολύ επεξηγηματικό και ε, περιγραφικό τρόπο. Θα δούμε ε, τι θα μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τους αριθμούς εγώ δεν τα πάω πάντα καλά όταν λέμε αριθμούς χωρίς να ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω, γιατί, πώς, ποιος, πότε κτλ. Είναι μεγάλη εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Ενέργεια, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον. Ποιος θέλει να μιλήσει, ο κύριος Σόν. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους κοιόδους εισηγητές, οι οποίοι έχουν συμβάλει τον, τα μάλλα στη συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Αναφέρατε αρκετούς αριθμούς. Ε, είπατε ότι κυκλοφορούν πολλοί αριθμοί, Πρόεδρε, ανώτατα όρια, συντελεστές, ε, οροφές. Όλοι αυτοί οι αριθμοί και το γεγονός ότι 7 επιτροπές ε, στο Κοινοβούλιο εξετάζουν ταυτόχρονα αυτό το το καθιστούν ιδιαίτερα περίπλοκο, ούτως ή άλλως. Όμως εγώ θα επικεντρωθώ σε τέσσερα κέρια σημεία, το τα όρια, τους συντελεστές, τα καύσιμα και το 2020. Για το ανώτατο όριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το ανώτατο όριο του 5% για τα καύσιμα πρώτης γενεάς είναι ισόρροπη πρόταση. Για διαφορετικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί συμβάλλει κατά μεγάλο μέρος στην αναχέτηση των επιπτώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ε, έμεση αλλαγή χρυσή γη. Και επειδή υποστηρίζεται και από τις υπάρχουσες επενδύσεις του 2011, η πραγματική κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 4,7% του συνόλου. Το να θέσουμε το όριο στο 5% θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό ε, μεταξύ του αντικτύπου ε, μετρίασης αναχέτησης και των τρεχουσών επενδύσεων όπως τις γνωρίζουμε οι οποίε θα συνεχιστούν με τι ε, υποβουλίε που ήδη έχουν ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή βιοκαυσίμων ούτω ή άλλω. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε ότι το όριο του 5% ήταν ο σωστός αριθμός Με τα σημερινά δεδομένα. Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε διορατικοί και να κοιτάζουμε στο μέλλον. Γι' αυτό προτείναμε να υπολογίσουμε το συντελεστή ε, στον συντελεστή Κάζη στην περίπτωση της υποβολής εκθέσεων και μόνον. Θα ήταν αρκετά ευνηδιαστικό να συμπεριληφθεί τώρα στην προσμέτρηση, αλλά τα επιστημονικά στοιχεία ήδη έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται και όταν θα έχουμε αρκετά πορίσματα θα μπορούσαμε να εισάγουμε τέτοια μοντέλα και σε άλλους τομείς πολιτικής μας. Και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό αυτό και σε συμφωνία με την αρχή υποζεή. Επίσης, η έμεση αλλαγή χρυσής γης δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε σαφώς αποκλήσεις. Διότι είναι τόσο διαφορετικές ε, οι συνεισφορές, η παραγωγικότητα, η συγκομιδή, τα λοιπάσματα, η ποιότητα των προϊόντων, όλα αυτά πρέπει να προσμετρηθούν. Δεν υπάρχει τρόπο ακριβού υπολογισμού σήμερα. Δεν υπάρχει τέλειο μοντέλο και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε και θεωρήσαμε ότι η χρήση τη μελέτη και το να βασιστούμε στη μελέτη ΕΦΠΡΙ ήταν ο καταλληλότερη προσέγγιση. Πολλοί ομιλητέ ανέφεραν τα καύσιμα δεύτερη γενεά και το θέμα που ανακύπτει με αυτά. Καλό θα ήταν να υπάρχει κάποιο είδου στόχο για τα καύσιμα αυτά. Θεωρούμε όμω ότι το να θέσουμε το όριο του 5% και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια θα αποτελεί μέρος της χρήσης μας ή τα μαγειρικά έλαια και τα ζωικά λύπη θα μας οδηγήσει σε μια ε, ισορροπία σε ένα μερίδιο του 2,5% από το 10% του συνόλου. Δεν είναι κακό αυτό ο στόχο για τα καύσιμα δεύτερη Νομίζουμε ότι ήδη συμπεριλαμβάνεται και δεν υπάρχει δική ανάγκη να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, ένα δευτερογενή, ξεχωριστό στόχο. Ταυτόχρονα όμω αναγνωρίζουμε την ανάγκη να προωθήσουμε και τα ε, αποθέματα ζωοτροφών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουμε άλλες πηγές όπως η λιματολάσπη ε, για την παραγωγή τέτοιου είδου καυσίμων. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη και αναπτύξαμε τη δημιουργία αυτών των αποθεματικών, τα οποία περιλαμβάνονται στα παραρτήματα τη πρόταση. Και εδώ χρησιμοποίησαμε συντελεστέ 2 και 4, δηλαδή τη διπλή, την τετραπλή προσμέτρηση, για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε και αυτά τα δυναμικά, τα αποθεματικά μάλλον, στην στον συνολικό υπολογισμό μα. Να τη σκεφτήκαμε λοιπόν για τα καύσιμα δεύτερη γενιά. Πολύ από τους παρεμβαίνοντες ανέφεραν και το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές σήμερα χρησιμοποιείται στα τρένα, στους σιδηροδρόμους. Δεν βλέπουμε λόγο, το λόγο να το ενθαρρύνουμε αυτό έτσι περαιτέρω. ιδίω για τα αυτοκίνητα συμπεριλαμβάνεται στη νομοθεσία μας και αυτό μπορεί κανείς να το προωθήσει ω έχει για να υπάρξει χρήση περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στα αυτοκίνητα. Πολλοί αποσιώπησαν το τι θα συμβεί μετά το 2020. Μάλλον μα κατηγόρησαν ότι αποσιώπουμε το τι θα συμβεί μετά το 2020. Υπάρχει ήδη ένα πρώτο στόχο για το 2020 και επίτηδε κι εμεί ε, δεν ε, τοποθετηθήκαμε σχετικά. Πάντω, αν διαβάσετε την ιδεολογική έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλέ ιδεολογικέ σκέψει και ρήτρε αναθεώρηση και τι δείτε και με προσοχή, θα δείτε ότι είμαστε αρκετά ε, ακριβεί στη διατύπωση. Δεν θέλουμε επιπλέον επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις για τα ε, βιοκάψιμα μετά το σύστημα που έχει προβλεφθεί στο 2020, ούτε Και θα δούμε μέλλον κατά πόσον οι συντελεστέ ILOC μπορούν να συμπεριληφθούν στα κριτήρια εφορία στο μέλλον. Όμως θα τα κοιτάξουμε αυτά σε ένα υποθετικό σενάριο για το τι θα συμβεί μετά το 2020. Τα βασικά πολιτικά σημεία που πρέπει να σκεφτούμε σήμερα για το ανώτατο είναι το ανώτατο όριο, έφτατα κάσουμε δεύτερη γενέας και οπωσδήποτε περιμένουμε να ξεκινήσουμε με την εισηγήτρια και τους κοιόδους εισηγητές τις προσεχείς εβδομάδες ε, εντατικές διαβουλεύσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία ε, στην Επιτροπή σας τον μήνα Ιούλιο και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια αργότερα. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Äh, Ευχαριστούμε. Δεν εννοούσα απλώ ότι ασχολείστε με το περιβάλλον αλλά και με την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Τώρα καλωσορίζω μια αντιπροσωπεία του Σουηδικού Κοινοβουλίου και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια Λεπάζ για να καταλήξει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Όντως, θα επιθυμούσα για εγώ να καταλήξουμε σε ένα κείμενο με συμβαστικές λύσεις που να είναι ισόρροπο. Δεν θα απαντήσω σε κάθε μια από τις ξεχωριστές παρατηρήσεις και τα σχόλια. κατέγραψα όλ, όλα αυτά που άκουσα με λεπτομέρειες, άκουσα προσεκτικά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι θα πετύχουμε συμφωνία και για το ανώτατο όριο και για τους δευτερογενείς στόχους και να πω στην κυρία Γκροστέτ ότι τα ανέφερα τα θήκια προηγουμένως γιατί όντως πιστεύω ότι είναι μια τεχνολογική λύση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα να ληφθεί λοιπόν όντως υπόψη στον υπολογισμό των συντελεστών. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά σημεία όπου οι απόψεις μπορεί να συγκλίνουν, φάνηκε από όσα είπαν εμένα και η ΔΕ, και πιστεύω ότι πραγματικά στην επόμενη συνάντηση των συνοριξικεδών θα καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις, ώστε να μην έχουμε 500 τροπολογίες όταν ψηφίσουμε τον Ιούλιο μπροστά μας, θα έχουμε πιστεύω μια θέση ε, σταθερή, ισόρροπη αλλά και αρκετά ε, τολμηρή από την άποψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος ώστε να φανεί ότι έχουμε άποψη και θέλουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών πράγμα που ελπίζουμε να στηρίξουν και οι συνάδελφοι στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Κορίνα για αυτά τα ενθαρρυντικά σου λόγια. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετέσχουν. Στις 10 Ιουλίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Προχωρούμε στο σημείο 14 της ημερησίας διάταξης. Τροποποίηση οδηγία σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον εισηγητής είναι ο κύριος Ανδρέα Ζανώνη, στον οποίο δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα είναι και, και αυτό το θέμα, μάλλον είναι πολύ περιπλοκό. Μιλάμε για την οδηγία για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Οπότε θα ήθελα να μου αφιερώσετε κάποιο παραπάνω χρόνο, γιατί το θέμα είναι πραγματικά ευρύ. Στο σχέδιο έκθεσης που υπέβαλα στις 6 Μαΐου, Έβαλα πάνω, έλαβα πάνω από 200 τροπολογίε από τους συναδέλφου. Και εδώ θα προσθέσουμε και τι τροπολογίε που θα φτάσουν από τι επιτροπέ ΠΕΤΗ και ΤΡΑΝ, μεταφορών και αναφορών. Δεν θα σταθώ σε όλε τι τροπολογίε λόγω περιορισμού χρονικού, αλλά τα βασικά σημεία προβληματισμού. Εκεί που έχουμε τι περισσότερε τροπολογίε. Αυτό είναι οι εξαιρέσει, η συντονισμένη προσέγγιση, η ενιαία θηρίδα, το one stop shop όπως λέγεται, όπου εκεί θα πρέπει να δούμε τι σοβαρές επιπτώσεις υπάρχουν. Το screening επίσης, η συμμετοχή του κοινού, η απόφαση για την ε, χορήγηση αδειών και το σχιστολιστικό, φυσικό αέριο. Ε, εδώ οι σκιώδεις εισηγητές, Αρσένης, Φερέιρα και Μπελιέ πιστεύω ότι θα μπορέσουν στη συζήτηση που θα έχουμε να εμπλουτίσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με νέα στοιχεία. Έτσι πιστεύω ότι με τα στοιχεία αυτά θα καταλήξουμε σε μια αρίστη πρόταση. Λόγου χάρη για, τα, για, τις, ε, για τους προστατευόμενους ιστορικούς τόπου σε αστικά κέντρα πολιτιστικής κληρονομιάς του συναδέλφου Γκουτιέρες, αλλά και για τα σημεία για τα οποία ενδιαφέρεται το κοινό, με την ε, παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών, όπως πρότεινε ο συνάδελφος Αρσένης, και αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά και, το, και οι προσπάθειες απλούστευσης της διαδικασίας. Όσο για το εφικτό των κανόνων και την ιδιαιτερότητα του κάθε προγράμματος αλλά και το πώς εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να μου πει τι άποψη έχει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τροπολογίες της συναδέλφου Μπελιέ που θέλουν να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και τη συμμετοχή του κοινού αλλά και σε αυτές του συναδέλφου Φερέιρα που ζητά επανειλημμένος μαζί με τη συνάδελφο Κλάς να λάβουμε υπόψη και τον αντίκτυπο που θα έχει αρχικά ένα σχέδιο για, άλλους τροπολογ... για άλλες τροπολογίες από τους συναδέλφους ε, του ΕΛΚ αλλά και άλλους συναδέλφους όπως του, του κυρίου Κράμερ και Ντέβις και του κυρίου Στίβενσον εδώ υιοθετείται μια διαφορετική σκοπιά. Οι τροπολογίε αυτέ ε, επικρίνουν περισσότερο τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σκοπό έχουν να ε, ελαφρύνουν την δομή συνολικά τη οδηγία, διαγράφοντα και ορισμένα σημεία του κειμένου. Σκοπό είναι να υπάρξει περισσότερη ευελιξία στην όλη διαδικασία. Πέραν αυτών των παραχωρήσεων, νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι επιδιώκουν τον ίδιο κοινό στόχο να έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα πριν από το τέλο τη θητεία, ώστε να έχει στα χέρια τη η ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να επιτύχει του στόχου του 21ου αιώνα. Θα πρέπει μόνο να, προσέξουμε, να προσέξουμε να μην γίνει ένα βήμα ε, οπισθοχώρησης ουσιαστικά ε, στην πρόοδο που θέλουμε να επιτύχουμε και αυτό με καποιε τοπολογιε συναδελφών σε κέρια σημεία τη προταση Ο στοχο είναι να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων ώστε να υπάρξει ευρεία συμφωνία και μετά την καλοκαιρινή διακοπή να ξεκινήσουν οι συνομιλίες με την Λιθουανική Προεδρία από Σεπτέμβριο και να καταλήξουμε σε γρήγορη έγκριση της οδηγίας. Ειδού η ανάλυση των βασικών προβληματισμών, βάσει των οποίων ε, διατύπωσα και εγώ κάποιε συμβαστικέ λύσει, τι οποίε υποβάλλει στην κρίση των σκιωδών εισηγητών. Να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τις για τις διαλύσεις. Ε, υπάρχει εδώ απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όμως ε, η νομολογία αυτή προκαλεί και κάποια σύγχυση. Υπάρχει σχετική ασάφεια. Διότι όλα τα έργα διάλυσης ε, το θέμα είναι πώς θα γίνει ο συσχετισμός μεταξύ της διάλυσης τριών και σχέδι. Εδώ μιλάω για τι τροπολογίε Φλόρεν Κράμερ και τι υπόλοιπε. Αλλά και άλλοι συναδέλφοι όπω ο κ. Ασένη, αλλά και οι συνάδελφο Τίσεν, ο συνάδελφο Τίσεν, προτείνει στι κατεδαφίσει να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα σχέδια που αναφέρονται στα, στα παρατήματα 1 και 2. Εκεί δηλαδή που μπορεί να υπάρξει σοβαρό αντίκτυπο για το περιβάλλον. Στο κείμενο αυτό θα συμπεριλαμβάνονται Ενδεχομένω τροπολογίε, γκουτιέρε και αρσένε, τι οποίε εγκρίνω. Και αναφέρονται και στι καταθέσει βάσει του παρατήματος 4. Για την ενιαία θηρίδα, το One Stop Shop, Όπω λέγεται, με την συντονισμένη προσέγγιση και το ενιαία θηρίδα, γενικά πρέπει να πω ότι ήμουν ευνοϊκά διακείμενο. Λόγω τη απλούστευση διαδικασιών, την θέσπιση μια ενιαία αρχή ώστε να γίνει πιο ταχεία η εξέταση των αιτήσεων. Δεν θίξαμε λοιπόν τα σχετικά σημεία από την Ευρωπαϊ... πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν και υπήρξαν συγκεκριμένε αντιρρήσει από ομοσπονδιακά κράτη που θεωρούν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει ελεύθερα να επιλέγουν τη διοικητική διαδικασία που θεωρούν ε, την πλέον εύστοχη στο εσωτερικό τους και ότι η κεντρική αρχή θα πρέπει να τους επιτρέπει ελεύθερα να επιλέγουν. Αυτό όμως που περισχύει είναι να επιδιώξουμε τους στόχους της πρότασης, δηλαδή να συγκεντρώμε πληροφορίες για την ποιότητα του περιβαλλοντικού αντικτύπου ενός έργου. Πρωτού λάβουμε αποφάσεις τεκμηριωμένες. Οι τροπολογίε των συναδέλφων λοιπόν θέλουν η ενιαία θηρίδα να γίνει προοριτική. Το γεγονός ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος προκύπτει από το πεδίο εφαρμογή διαφορετικών οδηγιών θα πρέπει να σε οδηγήσει παρόλα αυτά σε ένα κοινό στόχο. Εκτός και αν τα κράτη-μέλη θεωρήσουν ότι η εφαρμογή τέτοιων διαδικασιών είναι δυσανάλογη, μπορεί να ζημιώνει τους στόχους που έχουν καθοριστεί. Παρομοίως, τα κράτη-μέλη που θέλουν θα μπορούν να διορίσουν υπεύθυνοι αρχή ώστε να διευκολύνουν την διαδικασία έγκρισης κάθε έργου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατυπώσει κατευθυντήρες γραμμές απαραίτητες για την θέσπιση και την υλοποίηση τέτοιων κοινών συντονισμένων διαδικασιών, που μπορεί να είναι και προαιρετικές. Ελπίζω να στηρίξουν οι συνάδελφοι αυτή την πρότασή μου. Για τους περιβαλλοντικούς παράγοντε Άλλο θέμα. Εδώ δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή από του συναδέλφου στο νέο κατάλογο των περιβαλλοντικών παραγόντων, βάσει των οποίων θα αξιολογείται ο αντίκτυπο ενό συγκεκριμένου έργου. Ιδίω οι κλιματικέ αλλαγέ. Εδώ κάποιοι συνάδελφοι πρότειναν νέο ορισμό της διαπικιλότητας βάσει της σύμβασης του ΟΗΕ ή τη διαγραφή τη. Ή την αναφορά της Φλωρίδας και της Πανίδας μόνο στο κείμενο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει η τιμνία τη επικοινότητα. Μιλάμε για οδηγία αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Όμω, το πώ θα διατυπωθεί ο ορισμό και όπω την πρότεινα εγώ, σκοπό έχει να διευκρινίσει τι εννοούμε με τον όρο αυτό. Δεν νομίζω ότι εδώ πάντω ε, διασκεδάστηκαν οι αμφιβολίε πολλών συναδέλφων. Οι σκιώδει εισηγητέ πρότειναν έναν ορισμό απλούστερο, ώστε να πούμε ότι η βιοπικιλότητα καλύπτει όλε τι διαστάσει τη χλωρίδα και πανίδα, όπω αρχικά είχε προτείνει η συνάδελφο Τίσα. Για του περιβαλλοντικού παράγοντε, σημαντικό φάνηκε να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το υπέδαφο, όπω είπε η συνάδελφο Μπέλιε, ενώ είδα και την τροπολογία του κυρίου Στίβενσο σχετικά σε σχέση με τι καταστροφικέ συνέπειε. Για τι άλλε τροπολογίε θεωρώ ότι αυτέ που αφορούν τι κλιματικέ αλλαγέ ήταν πολυάριθμες και αντιφατικές. Θεωρώ ότι οι τροπολογίες Φλόρενς, Σόνικ, Σίμπερ και Στίβενσον που ζητούν τη διαγραφή του όρου αλλαγή επιτρέπουν να λαμβάνεται υπόψη παράγοντα επιρροή του κλίματο. Επειδή παρόλα αυτά είναι ε, σαφής η θέλησή μου να καταπολεμηθούν ε, όλες οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει στη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπο ενό συγκεκριμένου έργου σε σχέση με το τοπικό κλίμα. Δεν είναι τόσο εύκολο υπολογιστή οι επιπτώσει σε σχέση με ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Ένα άλλο θέμα είναι το screening. Έχουμε το άρθρο 4. Το ενίσχυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνοντα ένα παράρτημα, το δεύτερο, με ε, παράλληλες προτάσεις που θα πρέπει να γίνονται προς την αρμόδια αρχή. Και εδώ προσυπέγραψα γιατί πολλοί συνάδελφοι θεώρησαν υπερβολική την υποχρέωση πληροφόρησης από την πλευρά του υποβάλλοντος το έργο σε ταυτόχρονο στάδιο. Εδώ θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να πλουστεύσουμε και να διευκολύνουμε το διάλογο μεταξύ αρμόδιας αρχής και αρμόδιου φορέα, διότι σε αυτή τη φάση πάντοτε υπάρχει ασάφεια και βεβαιότητα. Δεν συμμερίζομαι τι ροσπαστικότερε απόψει συναδέλφων που ζητούν την απλή διαγραφή του παρατήματο, όπω η Φλόρεν, Κράμερ και άλλοι, αλλά θέμουν επιρρεπέστερο στο να διατηρηθεί το παράρτημα 2α. Ώστε να μην ξεχνάμε ότι πληροφορίε που θα πρέπει να παρέχονται θα πρέπει να περιορίζονται σε συνοπτικέ πληροφορίε και στοιχεία, συνοπτικά στοιχεία, ώστε να μπορεί η αρμόδια αρχή να λάβει μια τεκμηριωμένη ε, απόφαση. Ελπίζω ότι η προσέγγιση αυτή θα συγκεντρώσει την στήριξη των συναδέλφων. Τι προσεχεί ημέρε θα μοιράσω και άλλε συμβουλευτικέ προτάσει που αφορούν άλλα πολύ ευαίσθητα σημεία τη ε, πρότασης. Πρώτα απ' όλα το σκόπινγκ. Όπως ξέρετε αυτό έχει να κάνει με τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομεριών που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο σχέδιο και την πρόταση σχεδίου όπως υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή. Οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ προκαλέσαν πολλέ φιλονικίε. Ζήτησαν απλούστευση τη οδηγία κάποιοι συνάδελφοι. Ενώ είμαι αντίθετο με το επίπεδο ευελιξία που ζητούν κάποιοι για την όλη διαδικασία. Η συντόμευση του χρόνου είναι ένα σημαντικό παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την επιτεύξη του έργου της αρμόδιας αρχής. Ω προ το screening, ήμουν υπέρ τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πιο άλλη προσέγγιση και θα είμαι υπέρ των τοπολογίων των συναδέλφων που οδεύουν προ αυτή την κατεύθυνση. Για την υποχρεωτικότητα του scoping. Είμαστε υπέρ αρκεί να διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται μόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά όταν ο υποβάλλον το απαιτεί ή όταν η αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αρχών, το θεωρούν αναγκαίο. προκειμένου να υπάρχει έλεγχο για την ποιότητα πληροφοριών σε σχέση με το υπερβολικό αντίκτυπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προστρέχει σε ε, εγκεκριμένου εμπειρογνώμονε για την περιβαλλοντική έκθεση, την περιβαλλοντική επαλήθευση. Αυτέ είναι δύο φάσει. Για να επιτευχθεί ο στόχο, όπω αναφέρω το σχέδιο έκθεση, θεωρώ, μαζί με άλλου συναδέλφου, ότι η εφαρμογή ενό τέτοιου συστήματο θα είναι και περίπλοκη και ε, ιδιαίτερα θα Ο ρόλος πιστοποίηση λόγου χάρη σε πολλά κράτη-μέλη, όπως τη δική μου την Ιταλία, ε, παραπέμπει σε συγκεκριμένε διαδικασίες και πολλές φορέ σε ιδιαίτερο γραφειοκρατικό άχθος. Γι' αυτό στην εκθεσή μου προτείνω τη διαγραφή τη πιστοποίηση, διευκρινίζοντας ότι ο υποβάλλον θα μπορεί να ε, ανατρέξει και σε εξωτερικούς συνεργάτες για τη σύνταξη της υπερβολικής έκθεσης. Αυτή βεβαίω δεν μπορεί να είναι πλούσια. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από αυτή την εταιρεία. Μάλλον δεν θα μπορούν να είναι ανεξάρτητοι από την εταιρεία γιατί θα είναι εσωτερική. Αλλά θα πρέπει να είναι αρμόδιοι, όπω είπε ο συνάδελφο Στίβενσον. Άλλα δύο λεπτά σα παρακαλώ και θα ολοκληρώσω. Α, ναι, ναι, Το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η αρμόδια αρχή πρέπει να μπορεί να επαληθεύσει το περιβαλλοντικό αντίκτυπο μέσω τεχνικών αρμοδίων εμπειρογνωμόνων ε, με τα ανάλογα προσόντα και αμερόληπτων ουδέτερων, ώστε επιστημονικά να προσφέρουν αντικειμενικές πληροφορίες Και ως προς αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε ή το ένα ή το άλλο. Εγώ θα έλεγα ότι μεταξύ των δύο ας διαλέξουμε αυτό με αυτές τι συγκεκριμένε διευκρινήσει. Και τα τελευταία τρία σημεία εξαιρέσει. Ο συνάδελφος Αρσένη αλλά και συνάδελφος Μπελιέ πρότειναν και ε, επεσήμαναν ότι αποτελεί υποβάθμιση της νομοθεσίας και των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η θέση των εξαιρέσεων. Για σκοπούς εθνικής ε, άμυνας όμως μπορεί να ε, χρησιμοποιηθούν οι εξαιρέσεις ή για τις περιπτώσεις της παρακολούθησης. Υπήρξαν πολλές τροπολογίες αντιφατικές εδώ. Και θα φροντίσω να αποβάλω συμβαστική τροπολογία σχετικά. Αντιτίθεμαι σε κάποιες από τις τροπολογίες βέβαια, διαφωνώ για αυτού που ζητούν την διαγραφή τη παρακολούθηση, καθώ οι αρμόδιες αρχέ μπορούν να εγκρίνουν ένα σχέδιο που θα έχει συγκεκριμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνονται βεβαίω μέτρα παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων. Εάν φανεί ότι υπάρχουν αρνητικέ συνέπειες από αυτή την μέτρηση, θα πρέπει να ληφθούν σχετικά μέτρα και διορθωτικές δράσει, όπω ζήτησε ο συνάδελφο Αρσένη, του οποίου την τροπολογία προσυπογράφω. Ολοκληρώνω. 60 δευτερόλεπτα αν επιτρέπετε για την αναδρομική ισχύ. Εδώ υπάρχουν πολλές τροπολογίες, παρόλο που περιθώριο ελιγμού για συμβαστικές λύσεις μπορεί να βρεθεί ε, για να καλυφθούν οι ανησυχίες των συναδέλφων, ώστε να υπάρχει και νομική ασφάλεια. Εδώ πρότεινα κάποια χρονικά όρια για να λάβουμε υπόψη την ε, πρώτερη υποβολή της ε, περιβαλλοντικής έκθεσης για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Θεωρώ εδώ τις σχετικές τροπολογίες δεν επιτρέπουν να βρεθεί συμβαστική λύση, διότι πραγματικά υπάρχουν ε, αποκλίνουσες απόψεις. Πάντως, του συναδέλφου Ντρότ Μπελιέ, τις τροπολογίες θα ζητήσω να γίνουν δεκτές οι τροπολογίε, εφόσον μιλάμε για την εξόρυξη χωρί να θίγονται οι υδρολογικοί παράγοντε, και μόνο τέτοια σχέδια να εγκρίνονται. Κλείνω λέγοντα ότι στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών στι 2.30 στι 25 Ιουνίου ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει. ώστε στι 4 Ιουλίου στο Στρασβούργο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση και να περάσουμε με διαπραγματευτική εντολή σε τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ τώρα να ακούσω τα σχόλια των σχεδόν εισηγητών και των υπόλοιπων συναδέλφων προ το Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Τώρα μας παρουσιάσετε 600 τροπολογίες. Μια τεράστια επισκόπηση κάνατε. Μπορείτε και ε, Κατηδία να τα δείτε αυτά με τους και ηγητές. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες εδώ. Το λόγο έχουν οι σκιώδεις από το ΕΛΚ πρώτη Κριστίνα Κουτιέρες. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά στις ομάδες, συμφωνήσαμε σε πολλά και οι προτάσεις μου σε μεγάλο βαθμό εισακούστηκαν από ό,τι φαίνεται. Αποτέλεσμα ότι πολλές φορές έχουμε κάνει κοινέ τροπολογίες. Για μένα ποια είναι τα πιο σημαντικά. Πρώτον, πρώτα θα πω τα κακά και μετά τα καλά. Η οδηγία αυτή μου φαίνεται ότι θέλει να αλλάξει λίγα. Αλλά μακροπρόθεσμα τι κάνει. Επανέρχεται στο τεράστιο βάρος που υπάρχει πολλές φορές ε, στη γραφειοκρατία. Αναπτύσσεται τεράστια γραφειοκρατία και αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες και αυτονομείται. Καμιά φορά είναι ενδιαφέρουσες, αλλά άλλοτε όχι. Και δεν καταβαίνουμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν χρειάζεται να κάνουν μελέτη αντικτύπου περιβαλλοντικού, γιατί αυτά είναι λιμένα πράγματα, δεν χρειάζεται κάθε φορά από την αρχή. Ποια ήταν η δική μου δουλειά, να βρω ε, περισσότερη απλούστευση και πολύ περισσότερη τυποποίηση. Απλούστευση για ποιο λόγο. Είναι ένας άξονας που είναι και στον ορίζοντα για την Ευρώπη 2020. Υπάρχουν οδηγίες για την απλούστευση και εκπλήσω με που το έγγραφο δεν λέει τίποτα για απλούστευση. Είναι πολύ απλό να απλουστεύεις και σε γραφειοκρατικό επίπεδο. Θα καταργήσουμε εκθέσεις περιτές πολλές φορές, ε, πιο μικρές προθεσμίες Γιατί πολύ συχνά σπάμε την ενιαία αγορά με τέτοιε προθεσμίες που δίνουμε σε διοικήσει για να απαντήσουν ε, και έχω κάνει και μια τροπολογία για την απλούστευση. Ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να δεχθούν τη συμβουλή επιτέλους να σταματήσουν ε, και να απλουστεύσουν τα πράγματα. Το παράρτημα. Γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Ας πούμε, η βιομηχανία τροφίμων όταν έχει εγκριθεί από ένα δήμο, από μια περιφέρεια, να ε, δουλέψει κάπου ένα εργοστάσιο, υποτίθεται ότι έχει φως, νερό, τηλέφωνο, δεν πειράζει το περιβάλλον κτλ. Και πολλές φορές είναι ντόπιοι αυτοί που δίνουν τις άδειε. Τώρα τι χρειάζεται να το επιβαρύνουμε κάθε φορά. Και είναι και πολύ καθαρές πολλές φορές αυτές οι βιομηχανίες. Χρειάζεται πολύ μεγάλη απλούστευση. Στη συνέχεια, το θέμα της τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορισμό υπέρ της ενιαίας αγοράς, αλλά είναι στη διακριτική ευκαιρία των κρατών να την εφαρμόσουν ή όχι. Α, πολύ ωραία. Τους λέμε, σας παρακαλούμε κύριοι, μπορείτε να την τυποποιήσετε. Γιατί όταν υπάρχει ένας κινητήρας Renault, Mercedes, ξέρω εγώ, που έχει πιστοποιηθεί, κυκλοφορεί σε όλη την Ευρώπη. Τώρα πολλές φορές πιέζουμε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και ζητάμε εκθέσεις που δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γιατί είναι αμυγός βιομηχανικές. Παλιά μιλούσαμε για τη βιολογία ε, και για την ενέργεια, αλλά τώρα πολλές επιχειρήσεις έχουν εντάξει στη λειτουργία τους το περιβάλλον και το καθαρό ε, της λειτουργίας. Α πούμε, όταν βάζουμε ένα βιολογικό καθαρισμό, δεν θα πρέπει κάθε φορά να εξηγούμε τι είναι ο βιολογικό καθαρισμό. αν ρηπαίνει, αν δεν ρηπαίνει, αν χρειάζεται μελέτη. Ε, ξεπερνάει πάρα πολύ το επίπεδο της περιφέρειας αυτή η απέτηση που βάζουμε πολλές φορές. Χρειάζεται να γίνει μια προσπάθεια. στη Γερμανία πολλές φορές ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, να υπάρχει ένα πρώτο screening, συμβουλεύω, πολλές περιπτώσεις, σε μεγάλα έργα, ε, ένα screening ε, ε, και να λέμε ότι κοιτάξτε αυτό είναι βιώσιμο ή δεν είναι. Κοιτάξτε τι κάνετε με το περιβάλλον. Να μην υπάρχει τεράστια μελέτη αντικτύπου που είναι 700 σελίδες πολλές φορές. Ψυχή δεν τα διαβάζει αυτά και κανένας δεν τα καταλαβαίνει ακόμα και αν τα διαβάσει. Αν θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση, ας γίνει μια πρώτη εκτίμηση και μετά βλέπουμε. Ας πούμε, στο νότο του Ηνωμένου Βασιλείου προγραμματιζόταν ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος και είπανε όχι, θα γίνει πρώτα ένα μεγάλο έργο. Ε, απερίφθη, γιατί δεν το θέλαν το μεγάλο έργο, πάει και ο αυτοκινητόδρομος. Αυτό είναι ε, ε, ο πρώτερος έλεγχος του screening και θα μας έλυνε τα χέρια. Μετά υπάρχει και ένα χρονικό περιθώριο που πρέπει να ε, ε, υποβληθεί η έκθεση. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε τρία-τέσσερα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα χρονικό διάστημα, εμεί λίγο παραπάνω, αλλά όριο να υπάρχει. Και ο ρυθμό των σελίδων ε, θα πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι κατάχρηση. και πολλά περιτά έξοδα δημιουργούνται. Το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική κληρονομιά ανέκαθεν ήταν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στις οδηγίες. Αλλά τα κράτη-μέλη το εφάρμοζαν ανάλογα με τις συνθήκες τους. Άλλες με καταπληκτικό τρόπο, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, ε, Γερμανία, αλλά άλλες χώρες δεν το περιλαμβάνουν αυτό καν ως ιδέα. Άρα, χωρίς να είναι δεσμευτικό, σας παρακαλώ, όχι δεσμευτικό, μην περδευόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτιάχνει ένα κατάλογο ε, όπως το άρθρο 6 του Habitat, για το τι χρειαζόμαστε, έναν οδηγό να μας δώσει. Γιατί μετά έχουμε διάφορες αναφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν ασχολήθηκε με αυτά τα κριτήρια. Τελευταίο, που νομίζω ότι είναι και ενδιαφέρον. Η μεγάλη συζήτηση για την ενιαία αρχή. Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες που την έχουν αυτή την αρχή, έχουν έναν οργανισμό. Ε, αλλά και χώρες με περιφερειακή δομή δεν θα πρέπει να αλλάξουν. Αλλά δεν μπορούμε να καταδικάσουμε και μια χώρα που θέλει να έχει μια ενιαία αρχή να την αποκτά. Ε, για ε, το σκοπό της εναρμόνισης και της απλούστευσης. Λοιπόν, η σύσταση χωρίς να είναι δεσμευτικό να υπάρχει μια ενιαία αρχή, αν θέλεις. Και ένα τελευταίο επίμαχο και θέλω επιμείνω γιατί έχω ιδία πείρα από τη δουλειά μου. Εγώ δεν διαφωνώ. Καλά, το θέμα του εδάφους το έχουμε συζητήσει σε προηγούμενη έκθεση για τις ανανεώσιμες. Αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε μελέτη αντικτύπου σε συσπογενείς περιοχές ή σε παραποτάμια εδάφη, γιατί πλημμυρίζουν. Όλη η Ευρώπη έχει πλημμυρίσει. Και δεν είναι μόνο κλιματική αλλαγή, αλλά έχουν χτίσει τα ρέματα. Είναι σαφές αυτό. Ε, ε, να φτιάχνουμε αυτοκινητοδρόμους, αλλά τους έχουμε φτιάξει σε εδάφη που πλημμυρίζουν, σε μέρη που είχαν προβλεφτεί για να είναι λεκάνες απορροής και είναι αυτοκινητόδρομοι. Λοιπόν, στις όχθες των ποταμών θα πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα για περιοχές που να απορροφούν, να πλημμυρίζουν ε, εσκεμένα στη Γερμανία υπάρχει κίνδυνος ε, μεγαλύτερος ε, ε, πλημμυρών γιατί έχουν γεμίσει κανάλια τα ποτάμια. Και στις σεισμογενείς περιοχές δεν λέμε να μην χτίζονται, αλλά φαίνονται από πολλούς σεισμούς στην Ευρώπη ότι οι οδηγίες που δίνονται για την οικοδομή είναι πολύ διαφορετικές ανάλογα με τη σεισμικότητα του εδάφους. Λοιπόν, να πούμε, σε σεισμογενείς περιοχές θα πρέπει να έχετε ένα κανονισμό. Και τα σπίτια δεν πέφτουν όταν κάνει σεισμό εκεί, γιατί είναι αντισυσμικά. Καμία σχέση αυτό δεν έχει με την οδηγία για τη χρήση των γεών και τα εδάφη. Να μην μπερδευόμαστε. Αυτά ήταν τα γενικά που ήθελα να πω. Για μένα, απλούστευση, διευκόλυνση, λιγότερη γραφειοκρατία και τα λοιπά είναι εκ των όν ουκάνευ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Αρσένης, παρακαλώ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό νομοθέτημα αυτό που τροποποιούμε εδώ. Από το κύρια μελήματά μας θα πρέπει να είναι η ανεξαρτησία αυτών που θα κάνουν την μελέτη αξιολόγησης. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αδέκαστοι και ότι θα μπορέσουν να ταυτίσουν τα προβλήματα και να βρουν κάποια λύση, να κλείσουν παραθυράκια ή ελλείψεις παραθυράκια του νόμου που είχαν χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για να παραβιαστεί στην ουσία η εφαρμογή της νομοθεσίας πρέπει να γεφυρώσουμε κενά όπως για το πετρέλαιο και το αέριο κάνουμε τις αξιολογήσεις για κάθε εκμετάλλευση. Αλλά δεν γίνεται αξιολόγηση της έρευνας. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να είναι πιο σαφή, να είναι υποχρεωτική η αξιολόγηση. Τέλος, για την απλοποίηση και την αποσαφήνιση του υποχρεωτικού χαρακτήρα και τη καλύτερη πρόσβαση και πληροφόρηση του κοινού πρέπει να έχουμε ένα, μία ενιαία ιστοσελίδα σε κάθε χώρα. Μην είμαστε πια στη δεκαετία του 70 ή του 80 ή και στις αρχές του 90 όπου ο καθένας τα διάβαζε όλα στην εφημερίδα. Εμείς Ζούμε στην μεταιντερνετική εποχή. Whatever we do in the environmental impact assessments. Πρέπει λοιπόν σε ένα, σε μία και μόνη ιστοσελίδα. Και άλλα θέματα βέβαια αναφέρθηκαν από τον εισηγητή, αλλά αυτές είναι οι κύριες ιδέες. Ο εισηγητής χαρτογράφησε πολύ λεπτομεριακά τα θέματα σε έναν τυπούκητο των προβλημάτων και γι' αυτό αξίζει συγχαρητηρίων και ισχυώδης επίσης για την καλή συνεργασία από όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπελιέ από τους Φρυσίνους, παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα περάσω στην ουσία γιατί πολλά υπόθηκαν ήδη. Να ευχαριστήσω ξανά και εγώ τον εισηγητή, τον κύριο Τζανόνη, για την ποιότητα του έργου του από τη μια και για την ε, προθυμία του να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερομένους, όπως τα λέγαμε, για αυτή την αναθεώρηση οδηγίας για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο η πυγμή και η διάθεσή του να βρεθούν συμβαστικές λύσεις που να ικανοποιούν όλους μας απέτρεψαν να επιτελέσουμε ένα βήμα πρόοδου για να καλύψουμε τις ελλείψεις και τα κενά της υπάρχουσας νομοθεσίας. Αυτό ακριβώς ήταν και το αντικείμενο της προσπάθειας αναθεώρησης του κειμένου για τις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις. Πολλά, πολλές τοπολογίες έχουν υποβληθεί. Τις ε, σχολίασε ο εισηγητής, μεταξύ αυτών κάποιες είναι επικοδομητικές και εύστοχες. Πάντως, σε αυτή τη φάση θέλω να διαπιστώσω και να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι αρκετές από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν μόνο σκοπό είχαν να περιορίσουν το πεδίο της νομοθετικής πρότασης. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν αυτή ήταν η αρχική πρόθεσή τους, εάν όμως εγκριθούν αυτό θα γίνει, μπορεί μάλιστα να μας οδηγήσουν σε υπαναχώρηση σε σχέση με το ύψος επατήσεων της ε, σε νομοθεσία νομοθεσίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων ε, στο περιβάλλον. Κάποιες είναι πολύ σαφείς, ε, μακρο, διορατικές και λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιτρέποντας τις αρμόδιες αρχές να κάνουν τις σωστές επιλογές ώστε να επιλέξουν τα πλέον ισορροπά σχέδια και να προσφέρουν ε, ασφάλεια δικαίου στην περίπτωση που προκύψουν διαφορές μετά την έγκριση, επίσης να προστατεύσουν τη διαφάνεια και όλα αυτά σωστά μας τα θύμισε ο εισηγητής. Στόχος, σκοπός μάλλον είναι να επιδιώξουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020, για το Horizon 2020, μεταξύ των οποίων οι περιβαλλοντικές επιπτώσει και η καταπολέμηση των ε, κλιματικών αλλαγών καθώ και η υποβάθμιση τη βιοποικιλότητας. Νομίζω το χειρότερο θα ήταν να αποδυναμώσουμε του ισχύοντε κανόνε ε, σε σχέση και με την οικολογική κρίση που διανύουμε. Θα πρέπει να διατηρήσουμε αμύωτε τι φιλοδοξίε μα ω προ το στόχο του κειμένου και αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο οι τροπολογίε, οι συμβαστικέ τροπολογίε που είναι ο εισηγητή, στη φάση αυτή από την πλευρά, από τη σκοπιά της ομάδα των Πρασίνων μας βρίσκουν σύμφωνο, τη στηρίζουμε. Βέβαια αυτό θα το επαναλάβω και θα επιμείνω με μια απαγορευτική γραμμή. Ένα απαγορευτικό όριο. Αν αποδυναμωθεί το κείμενο όπως έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί θα στείλουμε ένα πολύ αρνητικό μήνυμα ως προς τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με το Συμβούλιο, αλλά και ιδιαίτερα αρνητικό προς τους πολίτες το σύνολο των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του οικονομικού χώρου θέλουν να συμμετάσχουν σε μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης οικονομίας. Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων επανειλημμένως από την αρχή της θητείας μας. Εάν λοιπόν υπαναχωρήσουμε ως προς τους στόχους αυτούς σε σχέση με το κείμενο, ε, θέτουμε ε, ένα βιβόλο, εν κινδύνο την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει ως τώρα. Και γι' αυτό θα στηρίξουμε τον εισηγητή ώστε να προωθηθεί η φιλόδοξη τοποθέτηση αυτή του Κοινοβουλίου και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να οδεύουμε στην κατεύθυνση των σωστών συμβαστικών λύσεων με μόνη μέρημνα το πνεύμα της νομοθεσίας αυτής και το αντικείμενό της να προστατευθούν και να τα έχουμε διαρκώς κατά νου στο επίπεδο των εργασιών μας. Είμαστε την Επιτροπή Περιβάλλοντος, όχι Βιομηχανίας, Θέλουμε μια συνολική ε, όμως ε, συμπερίληψη των περιβαλλοντικών στόχων στις επιλογές υποδομών που θα γίνουν, είτε για οικονομικούς είτε για μηχανικού σκοπούς. Κύριε Τζανόνι, λοιπόν, να υπολογίσετε στη στήριξή μας. Στην μέγιστη στήριξή μας. ώστε από το κείμενό σας, από την πρότασή σας, να προκύψει το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξιών και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ και για τη διαπίστωση ότι εδώ είμαστε Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να συζητάμε γενικότερα και να θέτουμε τις απόψεις μας και να τις φωτίζουμε. Ο κύριος Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Ζανώνη για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριέλαβε και τις απόψεις όλων των σκιωτών. Με εξέπληξε ο ρυθμός των τροπολογιών γιατί από τις πρώτες συναντήσεις που είχαμε το Μάιο όλοι οι σκιώδεις φαινόταν να υποστηρίζουν τις απόψεις του κύριου Ζανώνη. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό που τώρα έχουμε πάνω από 500 τροπολογίες. Βέβαια και εγώ ο ίδιος Έχω καταθέσει πολλές από αυτές. Ελπίζω να αντικατοπτρίζουν την πρόταση οδηγίας, όχι κανονισμού. Σωστά, γιατί στόχο έχουν οι τροπολογίες μου να επιτευχθεί η ευελιξία. Και αυτό κυρία Πρόεδρε δεν είναι προσπάθεια αποδυνάμωσης της αρχικής πρότασης της Κομισιόν, αλλά αναγνώριση του γεγονότος ότι σε μια εποχή λιτότητας δεν μπορούμε να επιβάλλουμε περισσότερη γραφειοκρατία στα κράτη-μέλη, αλλά ευελιξία. Είμαι λοιπόν απολύτως υπέρ αυστηρών ελέγχων και μέτρων αλλά πρέπει να διατηρείται η ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Τα κύρια θέματα βεβαίως είναι η εφαρμογή μιας συντονισμένης αξιολόγησης για το περιβάλλον και τη νέα διαδικασία screening και προσπάθησα να τα καλύψω όλα αυτά στις τροπολογίες μου. Στο άρθρο 2 υποστηρίζω την αρχή του One Stop Shop αλλά εθελοντικά πρέπει να αναγνωρίσουμε την ατομικότητα, τον ατομικό χαρακτήρα των οικονομικών σχεδίων και μελλοντικών σχεδιασμών της κάθε χώρας. Συμφωνώ απόλυτα με την Κομισιόν ότι για να αποφευχθεί η περίπτωση το screening να είναι υπερβολικά γενικό και είμαι κατά της εξάμηνης προθεσμίας για το screening. Τώρα για το υποχρεωτικό scoping στην 5 θέλω να συμπεριληφθούν όλα τα ιδέες που έχουν ακουστεί αλλά δεν είναι ρεαλιστικό να ζητούμε να πληροφορίες και για εναλλακτικέ λύσεις κάποιου που έχει αναλάβει το έργο, ο οποίος μπορεί να μην έχει αυτές τις πληροφορίες. Όπως ξέρετε τώρα η πιστοποίηση των ε, πυρογνωμόνων είναι σημαντικό τμήμα της οδηγίας και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όλες οι ΕΠΕ να γίνονται με αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό η φράση που προτιμώ αντί για διαπιστευμένη είναι σε αυτό που προτιμώ. Επίσης ξέρω ότι ο ορισμός της διαδικασίας διαπίστευσης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Και αυτό το ίδιο, καθε αυτό, θα μπορούσε να δημιουργήσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εκτός αυτών έχω υποβάλει και τροπολογίες για να υπάρξει μεγαλύτερη δημόσια συμμετοχή και να αναγνωριστεί ότι οι αρνητικές συνέπειες προς το περιβάλλον καμιά φορά καταλήγουν και σε αρνητικές συνέπειες και για την αξία της περιουσίας κάποιου που κατοικεί κοντά σε αυτά τα προγράμματα. Αυτό δεν το έχω δει να αναφέρεται αλλά είναι σημα... αλλού, αλλά είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και το συναντάω πολύ συχνά στην περιφέρειά μου ε, για τις συμβιβαστικές. Με ανησυχεί ιδιαίτερα κυρία Πρόεδρε το γεγονός ότι οι τύρφοι, οι περιφέρειες όπου υπάρχει τύρφοι έχουν σχεδόν καταστραφεί γιατί παράγεται πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα από εκεί αν καλλιεργηθεί. Και ήλπιζα αυτό να καλύπτεται από αυτά που λέει η πρόταση για τα εδάφη, για τις γέες. Αλλά πολλές χώρες μέλη όπως και η δική μου δεν θεωρούν την τύρφη ως έδαφος, ως χώμα, αλλά ως μέταλλο και θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν δεν καλύπτεται η τύρφη από τη γενική κατηγορία των γεών ή των εδαφών. Μπορεί να χρειαστεί λοιπόν προφορική τροπολογία ή προφορική συμβιβαστική τροπολογία, αλλά θέλω την πληροφορία. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Ζανώνη και όλους τους κοιότης για τη συνεργασία και ελπίζω να στηριχθούν οι τροπολογίες μου από την Επιτροπή ώστε να είναι καλύτερη η οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε με τους σκιώδεις ηγητές, τους παρόντες ε, μη τι άλλο, αλλά έχουν ζητήσει το λόγο τέσσερις ακόμα συνάδελφοι και θα μιλήσω κι εγώ αν προκάνω, αλλά επειδή η ώρα έχει προχωρήσει ε, κάπως ε, να αυτοπεριοριστούμε παρακαλώ. Ένα τρίλεπτο έκαστος, εντάξει. Ο Καλ Χάιντς Φλόρενς, παρακαλώ. Ε, σύντομος με χαρά, γιατί έχουν υποθεί πολλά ήδη. Η Κριστίνα Γκουτιέρες είπε ότι θα πρέπει να είναι πιο απλή η διαδικασία, λιγότερο κρατική. Ε, και να υπάρχει και προστιθέμενη αξία. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει διαβούλευση ε, με 2.004 απαντήσεις. Οι μισές από τη δική μου χώρα βέβαια. Και ρωτώ, για ποιο λόγο έγινε αυτό. Γιατί ακριβώς στη Γερμανία ε, βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας. Διότι το θέμα ποιο ήτανε. Η μεγαλύτερη δεύτερη εφαρμογή και τα προβλήματα συντονισμού είναι εκεί. Ε, και ερωτώ, αν τα κάνουμε όλα στην Ευρώπη ε, ισοπεδωμένα και ίσα, είναι πιο απλό. Το θέμα ότι έχουν οι Γερμανοί τόσα προβλήματα για μένα σημαίνει ότι φταίνει οι Γερμανοί. Δεν θέλω να μπω σε αυτό, αλλά ε, ε, αυτός ο χαρακτήρας ε, ο ίδιος της περιβαλλοντικής ε, μελέτης είναι προβληματικός. Είναι σαν να έχεις ένα κορμό και πας και κολλάς διάφορα χαρτιά. Δεν ξέρω μπορούμε να το εναρμονίσουμε στην Ευρώπη. Θα ήθελα να αφήσω στις περιφέρειες μια στοιχειώδη ευελιξία, βάση περιπτώσει. Βέβαια, κοινή μα στόχη θα πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστοί. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Έχω μεγάλε επιφυλάξει ω προ του εμπειρογνώμονε. Στη χώρα μου, Υπάρχουν και ειδικέ εγκαταστάσει ε, αυτοκίνητο, βιομηχανία, χημεία, πετρέλαια κτλ. Παντού. Αλλά για κάθε ειδικό εργοστάσιο χημίας θα πρέπει να ψάξεις και να υπάρχει ειδικό εμπειρογνώμων, τολμώ να το αμφισβητήσω. Υπάρχουν αρχές, υπάρχουν αυτοί που φτιάχνουν το εργοστάσιο, υπάρχουν ε, ε, εμπειρογνώμονες, πανεπιστήμια, αυτοί δεν μπορούν να συνεργαστούν για να φτάσουν σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι αυτή η ισοπαίδωση παντού των εμπειρογνωμόνων για τα πάντα, ε, και αυτό με κάνει να αμφιβάλλω. Και ανησυχώ λίγο ε, για την εναλλακτική εξέταση. Αν θέλω να φτιάξω ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο που δεν θέλω, ε, δεν θα ήταν σωστό πιστεύω εναλλακτικά να κοιτάξω αν χωράει και μια ανεμογεννήτρια. Γιατί έτσι θα πτωχεύσει από την αρχή η επιχείρηση. Αν έρχεται μια ε, περιφέρεια και πει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση που είναι ανεμογεννήτρια, να το κάνει. Αλλά όχι από την αρχή ο ίδιος ε, ο ενδιαφερόμενος να δεσμευτεί ότι θα έχει και εναλλακτική πρόταση. Έχω γράψει πολλά πράγματα, αλλά οι έξυπνοι συνάδελφοι με πρόλαβαν, με κάλυψαν και σταματώ, Πρόεδρε κοιτήρισε και το χρόνο σου. Μπράβο. Η Φρανσουά Κρουστέτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και οφείλω να σας πω ότι θα είμαι πολύ σκληρή στην τοποθέτησή μου διότι ανησυχώ βαθύτατα για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βγαίνουμε από μια οδηγία το 2009 που δεν έχει μεταφερθεί πλήρως σε πολλά κράτη-μέλη και πάλι μας προτείνουν ε, εκ νέου ένα καινούριο κείμενο. Πού να βρούμε τον μπούσουλα που έχουμε χάσει. Ε, θέλουμε να έχουμε καλή ε, μεταφορά μιας οδηγίας προτού περάσουμε στην επόμενη. Όποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εχουμε καλη μεταφορα μιας κείμενο λιγότερο δεσβάσταχτο και απλούστερο και πιο σαφές, ε, δεν το πετυχαίνει, ούτε αυτή τη φορά το πέτυχε. Εδώ λοιπόν η πρόταση είναι και επαφής και μακροσκελής και επιφέρει κόστος στην υλοποίηση και θα σας δώσω απλώς κάποια παραδείγματα. Εάν κοιτάξουμε καταλεπτό το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε ότι αν το κείμενο ε, υλοποιηθεί ω έχει, θα αυξηθεί το κόστο των βελετων κατα κατά 40-60%. Είναι η στιγμή για τέτοιου είδου επενδύσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσης η διαδικασία του screening, τα είπαμε και πριν, διερωτάται κανείς σε τι θα εξυπηρετήσει η υποχρέωση υλοποίηση μελε... εκπόνηση μελέτη αντικτύπου για να δούμε αν πρέπει όντω να γίνει μετά η κανονική μελέτη αντικτύπου. Άμα δει κανείς το κείμενο και τα παρατήματα, αρχίζει και λέει, σκέφτεται τι φρικτά πράγματα είναι αυτά που προτείνονται σε ό,τι αφορά τι προθεσμίε. Έγινε και λόγο για τι προθεσμίε εντό εισαγωγικών θέλαμε κάποιε λογικέ ε, προθεσμίε. Όμω εδώ και πάλι επικρατεί η ασάφεια. Δεν μπορούμε να ορίσουμε τι ε, περιμένουμε με ακριβεί προθεσμίε για κάθε στάδιο τη διαδικασία. Και δεν μπορούν να αποφευθούν ούτε καθυστερήσει για την ε, λήψη αποφάσεων για επενδύσει, ούτε το επιπλέον κόστο. Μιλάμε για σχέδια επενδύσεων, εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και λέμε θα χρειαστούν λογικές προθεσμίες έτσι γενικά και αόριστα. Δεν είναι, είναι αδιανόητο αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ ακριβεί για κάθε στάδιο τη διαδικασία. Ο ε, ορισμό του όρου βιοπικιλότητα είναι τελείω ασαφή κι αυτό από τη μια λέμε βιοπικιλότητα και από την άλλη ε, χλωρίδα και πανίδα. Μα υπάρχουν συγκεκριμένε περιοχέ, τα υπερπόδια διαμερίσματα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ε, πλήρω όλα τα ζωικά και φυτικά είδη που μπορεί να υπάρχουν και σε όλο το εύρο την βιοπικιλότητα αυτών των τόπων. Τι σχέδιο θα γίνει εκεί, τι επενδύσει, τίποτα. Δεν γίνεται κι αυτό. Και έπειτα το κερασάκι στην τούρτα είναι η υποχρέωση δημοσίευσης της πιθανής ε, ισχύουσας κατάστασης του περιβάλλοντος εν απουσία σχεδίων. Μα είναι τελείω ανέφικτο κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση, πού είναι τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα, οι αξιοσημείωτε επιπτώσει στο περιβάλλον, αν δεν υπάρχουν ούτε καν σχέδια προγραμμάτων. Σα τα λέω αυτά για να δείτε πόσο είναι όλα αυτά παράλογα. Δεν είναι λογικά τα πράγματα αυτά. Το άρθρο 3 ε, απαιτεί όλοι οι υποβάλλοντε σχέδιο ή οι συμμετέχοντε να υποβάλουν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν την μεταφορά τη αναθεωρημένη οδηγία για να συμμορφωθούν με τι ενδεχόμενε υποχρεώσει που θα προκύψουν να δεν έχει ολοκληρωθεί. Μα καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο μέτρο τι θα κάνει, θα πάυσει τι περισσότερε από τι ε, προσπάθειε που ήδη γίνονται και όλα τα σχέδια που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή και θα πάψουν όλα. Είναι η πλέον αρνητική θεώρηση τη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία ε, και και της δίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οι πολίτες δεν περιμένουν αυτά από εμά, κυρία Πρόεδρε. Περιμένουν ε, προβολή για τις μελέτες αντικτύπου. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη προβολή και διάδοση και βεβαίως χρειάζεται ε, προώθηση των σχετικών πρωτοβουλειών θα καταρρεύσουν τα τοπικά σχέδια και θα γίνουν ουσιαστικά μια φυλακή διοικητική και γραφειοκρατική. Ευχαριστώ, καλώς Jag vill säga att, ähm, vad skulle du säga du, Grostet, om det visar sig... Κυρία Γκροστέτ μου, τι θα λέγατε αν, αν λέγω, αν βρισκόταν ένα φάρμακο για τον καρκίνο με αντίτιμο λέει την κατάργηση των μελετών αντικτύπου για το περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα φάρμακα προέρχονται από φυτά και αν καταστραφεί το περιβάλλον θα χάσουμε πολύ περισσότερα από απλώς φυτά δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι λογικό να μην βγάλουμε συμπαράσματα από τις στρατιωτικές ας πούμε επενδύσεις οι οποίες οπωσδήποτε εφαρμόζονται. Υπάρχουν οι τροπολογίες των πρασίνων, θυμάστε ότι όταν συζητούσαμε το θέμα την προηγούμενη φορά θέλαμε να ρωτήσουμε σε τι βαθμό η βιομηχανική εκμετάλλευση καταλήγει σε μόλυνση με βαρέα μέταλλα. Χρειάζεται λοιπόν σε όλες τις περιπτώσεις που ανέφερα μελέτη αντικτύπου και να εξετάζονται και τα εναλλακτικά σχέδια να είναι υποχρεωτική εξέταση των εναλλακτικών. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στη δική μου χώρα και σε άλλες. Χρειάστηκε να εξεταστούν εναλλακτικά προγράμματα για τη διαδρομή κάποιου σιδηροδρόμου κλπ. Και ήταν θετικό αυτό. Χρειάζονται Χρειάζεται η εξέταση των εναλλακτικών. Αλλιώς ρίχνουμε, πετάμε τα λεφτά από τα παράθυρα και μετά χρειάζεται να διορθώσουμε τα αδιόρθωτα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Λέει ο κύριος Κράμερ, συμφωνώ με τον κύριο Φλόρεντς και με την κυρία Κροστέτ που το είπε με τόσο πάθος Ισχύει μια μελέτη αντικτύπου για το, ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εφαρμόζεται σωστά στα περισσότερα κράτη-μέλη. Και εγώ κατάγομαι από το ίδιο κράτος με το Φλόρεντς και ε, καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες να ε, υλοποιούμε ε, αυτή τη μελέτη όπως επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία. Αλλά εκεί που εφαρμόζεται και εφαρμόζεται καλά δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Λοιπόν, Αντί να αρχίσουμε να επεκτείνουμε την εφαρμογή και το πεδίο εφαρμογής, να φροντίσουμε καλύτερα να εφαρμόσετε σωστά εκεί που γίνεται ε, λοιπός η εφαρμογή της. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίκαιρο και καλό. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Το θέμα δεν είναι να ε, μειωθεί το περιβαλλοντικό δίκαιο, μην με παρεξηγήσετε παρακαλώ, ε, ούτε να είναι εις βάρος του περιβάλλοντος, αλλά τέτοιες ώρες τέτοια λόγια να κάνουμε προτάσεις για αλλαγή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπαίνει στο ίδιο το δίκαιο των διαδικασιών ε, για τα έργα. Φανταστείτε πόσο χρόνο θα χρειάζεται ένα έργο για να διοδοτηθεί, για να εγκριθεί. Η μελέτη αντικτύπων σημαίνει ότι εκ των προτέρων ε, εκτιμάς τι αντίκτυπο θα έχει στο περιβάλλον ένα έργο που θα γίνει στο μέλλον. Και υπάρχει και ένα ειδικό δίκαιο, ας πούμε, ε, η οδηγία για τη χλωρίδα και την πανίδα, η προστασία των πτηνών, ξέρω εγώ, και ένα σύνολο, ε, ένας όγκος άλλων νομοθετημάτων. Αυτό δεν θα πρέπει να προεξοφλείται από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι ένα δίκαιο που θα το βρει μπροστά του το έργο στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της έγκρισης και της αδειοδότησης. Δεν καταλαβαίνω τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το είπε και η κυρία Γκροστέτ και ο Καλχάιντς Χάιντς Φλόραντς. Ότι θα πρέπει η ίδια η αρχή, λέει, να αποφασίζει μια εναλλακτική πρόταση. Έρχεται ένας και θέλει να φτιάξει ένα, ας πούμε, θερμοελεκτρικό εργοστάσιο. Μπορεί η ίδια η αρχή, η αρμόδια, να του πει, σύμφωνα με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, α όχι δεν θα φτιάξει τέτοιο εργοστάσιο, θα πρέπει να κάνεις ε, άλλη τεχνολογία να χρησιμοποιήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ διευθυντικό και παρεμβατικό ε, βήμα. Και πού είναι η ελευθερία του επιχειρήν. Ούτε έχει καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχει ένα βασικό σενάριο για μηδενική βάση ότι θα πρέπει ο ανάδοχος να έρθει λέει να αποδείξει τι θα γίνει αν δεν γίνει το έργο του. Αυτό είναι η διαστροφή της ε, αφηρημένης έννοιας. Δηλαδή θα έλεγα να φτιάξω ένα εργοστάσιο και να έρθω να αποδείξω τι θα συμβεί αν δεν το φτιάξω το εργοστάσιο, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι καλή προστασία του περιβάλλοντος, ούτε σωστός τρόπος αυτός και φοβάμαι ότι στο τέλος δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εντάξει, καλό το περιβάλλον και η μελέτη περιβαλλοντικών αντικτύπων να διευρυνθεί, λέμε, αλλά και ταυτόχρονα να απλουστευτεί με λιγότερη γραφειοκρατία. Ε, αυτά τα δύο όμως δεν συνάδουν. Θα πρέπει να έχουμε μια μελέτη ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων που να διατηρεί το status quo. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να διευρυνθεί ε, ούτε αντικειμενικός ούτε κανένα άλλο. Αφήστε δε που και η αποδοχή αυτού του νόμου δεν θα αυξηθεί με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν μεταφραστούν όπως είναι σε νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα να πω και εγώ αυτά που ήθελα. Ακούστηκε μια δυσφορία και ε, συμφωνώ απολύτως. Ο Φλόρενς το είπε και ο Ρόμπερτ Κλάμε και ε, από τη Γερμανία και η κυρία Γκροστέτ παρουσίασε τη γαλλική θεώρηση. Μπορεί να ακούγεται απλό ότι θέλουμε άρση της γραφειοκρατίας, αλλά να ρυθμίζουμε τα πάντα μέχρι τελικής κεραίας. Μα πώς θα πάρει κάποιος άδεια ε, ε, ε, ή να υπάρχει κάποια δυνατότητα να χτιστεί, να δημιουργηθεί μια νέα εγκατάσταση. Δεν είναι μόνο αυτοκινητόδρομοι και σιδηρόδρομοι που χτίζουμε ή τρένα καινούρια ας πούμε φτιάχνουμε και σπίτια ακόμα, αλλά χρειαζόμαστε και ε, νέες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς θα φτιάξεις δίκτυο αν δεν μπορείς να κουνηθείς ούτε ρούπι. Και χρειάζεται μελέτη περιβάλλοντος και επιπτώσεων κτλ. Ε, και μέχρι τελευταία λεπτομέρεια και θα πρέπει να ασχολούμαστε και να είμαστε υποχρεωμένοι με την τελευταία λεπτομέρεια. Εγώ βλέπω στη χώρα μου μάλλον ότι όλοι αυτοί οι κανονισμοί και οι οδηγίες χρησιμοποιούνται για αποφυγή, αποτροπή. Και αν δεν ε, του περάσει κάποιο με την οδηγία για την προστασία των πτηνών, βρίσκει κάτι άλλο για την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Κάποιο που δεν θέλει να γίνει μια γέφυρα, ξέρετε δεχομένως το έργο στην περιφέρειά μου, το φρενάρι ε, ε, επικαλούμενος διάφορες οδηγίες και κανονισμούς. Α, και τώρα λέει, ελάτε να αποδείξετε τι θα γίνει αν δεν χτιστεί αυτή η γέφυρα. Δεν μπορούμε να ζητάμε και τον ουρανό με τα άστρα και άρση της γραφειοκρατίας. Ε, σαφή διαδικασία θέλουμε και ε, χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες σαφείς για τις άδειε και τις εγκρίσεις και θέλουμε να παίρνονται οι όχι να αποφεύγονται. Εγώ προέρχομαι από τη Γεωργία και έχω ένα καημό. Ε, κοιτάξτε πώς χρησιμοποιούνται σήμερα ε, ε, καλλιέργειες, οι αρρώσιμες γέες δεν τις αξιοποιούμε. Ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η χρήση των γεών. Δυστυχώς χάνονται από τις καλλιέργειες ε, και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα λάβει υπόψη της και σε συνένεση με τους ε, ενδιαφερμένους και τον εισηγητή να μπορέσει να τα προωθήσει όλα αυτά. Ο κύριος Κρεμλής τέλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας θυμίσω τον στόχο της πρότασής μας. Είναι διτός. Πρώτα απ' όλα να βελτιώσει την ποιότητα της διαδικασίας των ΕΠΕ και έπειτα να ευθυγραμμίσει την όλη διαδικασία ΕΠΕ όλα τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων του διοικητικού άχθους, του κόστους και των στοιχείων απλούστευσης, συζητήθηκαν όλα αυτά διεξοδικά με τη μελέτη αντικτύπου που παρήγαγε και εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα γνωρίζετε ότι ο υπεύθυνο της μελέτης αντικτύπου μας ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο και επιβεβαίωσε τα πορίσματα της μελέτης αυτής του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το φως αυτού του διτού στόχου που στην πρότασή μας είναι θεμελιώδου σημασίας και συμπεριλαμβάνει στοιχεία τα οποία πρέπει να συνεπάρξουν γιατί είναι αλληλοσυμπληρωματικά και κέρια, όπως είπα, σημασία στο πλαίσιο βελτίωσης του πεδίου της οδηγίας υπό το φως λοιπόν όλων αυτών των δεδομένων Εξετάσαμε τις υποβληθήσεις τροπολογίες. Τις ομοδοποιήσαμε σε δύο κατηγορίες. Τα σχόλιά μου θα αφορούν τις τρεις κατηγορίες που ανέφερε. Υπάρχουν τροπολογίες που επιδιώκουν περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάμωση της πρότασής μας, στηρίζουν τους στόχους μας, οπότε έχουμε μια καταρχήν θετική στάση απέναντί τους, αφορούν την ποιότητα των εκθέσεων ΕΠΕ, την ε, αποσαφήνιση των ε, χρονικών προθεσμίων και των επιλογικών σκέψεων ως προς την συλλογιστική των αναθεωρημένων ε, διατάξεων. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις τροπολογίες που στέκονται στο ύψος των στόχων της πρότασης, αλλά χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση για να αποσαφινιστούν κάποια στοιχεία τους. Να δώσω ένα παράδειγμα, κάτι που το ανέφερε και ο κύριος Τζανώνη, ε, τα έργα κατεδάφισης. Μπορεί να είναι μέρος ενός σχεδίου, οπότε θα πρέπει να εκτιμώνται και να αξιολογούνται ταυτόχρονα με το όλο το σχέδιο, συνολικά αλλά μπορεί να είναι και ένα αυτόνομο σχέδιο σε περίπτωση που κάποιος θα κατεδαφίσει ένα παλιό κτίριο, ε, τεράστιο κτίριο σοβιετικού τύπου, σε μια περιοχή που θέλει να δημιουργήσει μια πράσινη υποδομή. Στο κέντρο, ενός αστικού κέντρου. Αυτό, όπως είπε ο κ. Τζανόνι, θα πρέπει τουλάχιστον να περάσει από screening βάσει τη οδηγίες ΕΠΕ. Από την άλλη, συμμεριζόμαστε το στόχο αρκετών τροπολογιών για τον περιορισμό του πεδίου στις εξαιρέσεις. Αυτές είναι οι τροπολογίες 132, 33 και 160. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε θετικά διακείμενοι και ως προς την τυποποίηση που προτείνεται με την τροπολογία 189 με την προσθήκη της φράσεις η τυποποίηση θα μπορούσε να είναι ε, καλοδεχούμενη όπου είναι εύστοχη. Σε ό,τι αφορά την ε, πιστοποίηση των εμπειρογνωμόνων. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο όρος πιστοποίηση, accreditation, δεν είναι αποδεκτός ε, ομόφωνα. Εννοούμε εμπειρογνώμονες που έχουν την, ε, τα απαραίτητα τεχνικά και επαγγελματικά προσόντα, αποδεδειγμένη πείρα και μπορούν να διευκολύνουν στο έργο του τον υποβάλλοντα το, έργο, το, το σχέδιο. Έπειτα μας ενδιαφέρει το επίπεδο της εμπειρογνωμοσύνης των αρμοδίων αρχών, ώστε να μπορούν να εγκρίνουν και να αξιολογήσουν την ποιότητα του έργου όπως θα γίνει και στο επίπεδο του υποβάλλοντος και στο επίπεδο της αξιολόγησης από την αρμόδια αρχή. Άρα, επ' αυτού, θα μπορούσαμε να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση ώστε να πετύχουμε τον στόχο που από κοινού νομίζω επιδιώκουμε. The ε, third category, ε, Τρίτη κατηγορία, οι τροπολογίες που ξεπερνούν τα όρια της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είτε αναφέρονται σε διατάξεις που δεν κάλυψε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε στενεύουν τον κύκλο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ δυσκολεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τι αποδεχτεί. Γίνανε αναφορέ στην επικοινότητα τι κλιματικέ αλλαγέ και των κίνδυνων καταστροφών. Αυτέ είναι βασικέ προτεραιότητε και εν συντομία, όταν αναφερόμαστε εδώ στη Χλωρίδα και την Πανίδα, έχουμε υπόψη μα την οδηγία ε, βιοτόπων ε, οικοσυστημάτων μάλλον. Ε, η δική μας οδηγία είναι ευρύτερη. Υπάρχει λοιπόν επέ για τη βιοπικιλότητα και υπάρχει και εκτιμένο στη Γαλλία λόγω χάρη. Το όλο αυτό για την κυρία Γκροστέτ. Υπάρχει και εκτιμένο και προηγούμενο στη Γαλλία σε σχέση με εκτιμήσεις που γίνονται βάσει του γαλλικού δικαίου για την βιοπικιλότητα. Σε ό,τι αφορά το κλίμα, ο κύριος Τζανόνι αναφέρθηκε στην, ε, στον περίπλοκο χαρακτήρα ορισμό ενός σχεδίου που μπορεί να οδηγεί και να προκαλεί, να εντείνει τις κλιματικές αλλαγές. Κλίμα όμως δεν είναι μόνο το τοπικό κλίμα. Ένα σχέδιο μπορεί να έχει επιπτώσεις εκτός ε, τοπικών ορίων. Οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα φαινόμενο ευρύτερο, παγκόσμιο. Άρα αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να καλύπτεται από το σκόπινγκ. Μεταξύ άλλων πιστεύουμε ότι το scoping είναι μέθοδος ε, που θα είναι κέρια σημασία. Διότι θα επιτρέπει σε αυτό που βάλει το σχέδιο να δει τι ε, προκύπτει από τι νομικέ απαιτήσει και ποιε θα είναι επιπτώσεις επιπτώσει στην επικοινότητα ή παράγοντες κινδύνου. Σε πολλές περιπτώσεις η περιβαλλοντική έκθεση καλό είναι να μην έχει και ευρύτατο πεδίο, διότι ο αντίκτυπο μπορεί να είναι περιορισμένο. Οπότε το scoping είναι ένα εργαλείο χρησιμότατο. Και για, δώσω, αυτό που προτείνει το σχέδιο και γιατί θα είναι και ένα εργαλείο απλούστευσης για να αποφύγουμε περαιτέρω άχθος ή να πετάει τον μπαλάκι αρμόδια αρχή στον υποβάλλοντα και αντιστρόφως. Ή μετά να απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες από τον υποβάλλοντα σε κατοπινά στάδια της διαδικασίας και αυτό να εντείνει το κόστος και τη... να παρατείνει τη διαδικασία. Μια γενικότερη παρατήρηση τώρα που έχει να κάνει και με το σκόπινγκ. Ο κανονισμός 10 ή ε, για την ευθυγράμμιση των ΕΠΕ που έχουν εγκριθεί και προβλέπουν προθεσμίες για σχέδια κοινού συμφέροντας, προβλέπει υποχρεωτικό σκόπινγκ, υποχρεωτική ενιαία θηρίδα και υποχρεωτική αρμόδια αρχή είναι ήδη τμήμα του κεκτημένου μας, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κεκτημένου. Ο κανονισμός αυτός είναι μέρος της νομικής τάξης και της νομοθεσίας των κρατών μελών μας. Μιλάμε για μια διαδικασία ευθυγράμμιση που συνάδει και με την Ευρώπη 2020, τους στόχους δηλαδή τη θετικής αυτή. Όταν προτείναμε τον κανονισμό αυτό, ο σκοπός ήταν να επιταχύνουμε την έγκριση και τις παραγωγικέ εκτιμήσει με συντονισμένο ε, ενιαίο τρόπο για την προάσπιση κοινών συμφερόντων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασία. Επιτρέψτε μου να σας πω λόγου χάρη ότι στη Γερμανία, την Αυστρία και την Πολωνία, για να κατονομάσω μόνο τρία από τα κράτη-μέλη μας, έχουμε υποχρεωτικά κοινέ διαδικασίες. Η ενιαία θηρίδα λοιπόν ήδη είναι μέρος του δικαίου κάποιων των μελών. Πέραν των απαιτήσεων της οδηγίας και τώρα, ανέφερα το σκόπεν και πριν. Το σκόπεν είναι χρησιμότατο εργαλείο. Αισθανόμεθα ότι θα πρέπει να παραμείνει υποχρεωτικό. Εάν είναι δεσμευτική η χρήση του, θα εξυπηρετήσει και τον επαγάλλοντα και θα αποσαφηνίζει όλα τα στοιχεία περιβαλλοντικών πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται όπως τα προηγουμένως που έχουν να κάνουν προκότερα ζητήματα όπως το κλίμα, τη βιοπικιλότητα και το καθεξής, αλλά θα ορίζει και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε. Εφόσον η πρότασή μας δεν είναι να έχουμε μόνο δεσμευτική, κοινή, δεσμευτική, συντονισμένη διαδικασία, αλλά δίνει και τη δυνατότητα να έχουμε ένα συνδυασμό κοινών και συντονισμένων διαδικασιών. Σκεφτείτε τώρα, μπορεί να έχουμε κοινή ΕΠΕ βάσει τη οδηγία για του ε, οικοτόπου, για τα οικοσυστήματα και να συντονιστεί αυτό με άλλε οδηγίε όπω των υδάτων, ε, τις οδηγίες πλαίσιο, τη ΕΒΕΖΟ και ούτω καθεξής. Βέβαια οι πιο λογικές υπάρχουν λογικέ λογικές εναλλακτικές, αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Φλόρενς, οι οποίες έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο σχέδιο που υποβάλλεται. Η εξέταση των εναλλακτικών δεν θα οδηγήσουν στην απόρριψη και την ευθέτηση άλλου σχεδίου. Απλώς η εναλλακτική είναι να λέμε ότι δεν θέλουμε να το ονομάσουμε ε, επένδυση σε αυτό το τομέα, επένδυση στην αιωλική. Συγκεκριμένα για το σχέδιο που έχει εγκριθεί και για τις ε, ασφαλιστικές δικλείδες δεν καλύπτονταν από την πρότασή μας Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ιδίως όταν μιλάμε για την οριζόντια εξόριξη. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό στο επίπεδο του παρατήματος 1. Θα εξαρτηθεί βεβαίως από τα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται και από το πρόσθετο έργο που πρέπει να επιτελεστεί προκειμένου να διευκρινιστεί το πεδίο. Το πεδίο του τι τελικά θα και τι όχι. Ως προς αυτό πάντως να πω ότι είμαστε ανοιχτοί εφόσον οι δύο συνομοθέτες συμφωνήσουν. Και ακροτελεύτια παρατήρηση, τα εδάφη, τα οργανικά, η τύρφη. Κοιτάξτε, έχει τελειώσει ο χρόνο μας για σήμερα και ε, θέλω να δώσω το λόγο και στον εισηγητή. Αλλιώς θα μας φύγουν οι διερμηνείς γιατί σχολάνε. Ε, ο κύριος Τζανώνη. Είμαι πολύ συνοπτικός. Ευχαριστώ όλους για την υπομονή τους. Άκουσα με εξαιρετική προσοχή και ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους και εισηγητές και όσους πήραν το λόγο από την Επιτροπή για τη συνεισφορά τους. Και πραγματικά ανακουφίστηκα με τις παρεσβάσεις τους. Αν και κάπως ευνηδιάστηκα με μερικούς συναδέλφους, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι οι τροπολογίες μας οδεύουν σε σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε ένα κανόνα γιατί διανύουμε και περίοδο κρίσης και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, συγκεκριμένα πορεία που να ξέρουμε ότι θα ακολουθήσουμε με τρόπο σαφή. Και θα πρέπει να είναι και πιο εύκολη η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Να προσθέσω εδώ κάτι. Ακούγοντας κάποιες παρεμβάσεις, σκεφτόμουν καταστροφές που έχουν συμβεί στη δική μου την περιοχή. Πολλές χωματερές που έχουν ρηπάνει τους συντροφόρους ορίζοντας. Άλλες υποδομές που δεν έχουν οικοδομηθεί σωστά και προέκυψαν θύματα. Ή ε, καλλιέργειες σε λόφους που δημιουργήθηκαν για την καλλιέργεια και την παραγωγή προσέκο και τελικά κατέληξε να υπάρχει διολύστηση του εδάφους και να πληγούν οι γειτονικέ πόλεις στους πρόποδες. Πολλές περιπτώσεις με πολλά θύματα σε ανθρώπινες και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και οικονομικές επιπτώσεις που τις πολύ καλύπτουν συνήθως οι πολίτες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συνάδελφοι λοιπόν ανησυχούν αν ένα σχέδιο μπορεί να στοιχήσει 40-60% παραπάνω. με εφόσον εδώ μιλάμε για έργα που κρατούν 10-20-100 ε, χρόνια, όπως οι γέφυρες. Εδώ Αξίζει τον κόπο κάτι παραπάνω να το πληρώσουμε, να έχουμε προθεσμίες λίγο μεγαλύτερες και πιο αυστηρές, παρά στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστροφές οικονομικές, δυσανάλογες, απαράδεκτες και για τον επιπλέον λόγο ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις πόρους του πλανήτη και πρέπει να εφετήσουμε κανόνες που να μας λένε και να μας εξηγούν καλύτερα τι θα κάνουμε για να ετοιμάσουμε το πλανήτη και για τις μελλοντικέ γενιές. Ε, με όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα ε, θα ξανασυναντηθούμε ως, σε επίπεδο σχεδόν εισηγητών και θα αναζητήσουμε ε, με ένα σημείο ισορροπία και συμφωνία ώστε να προχωρήσει η εξέταση τη οδηγία αυτή και να καταλήξουμε με νέου κανόνε και σε συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, του ομιλητέ μα και του διερμηνεί ε, που ε, άντεξαν τόσες ώρες. Λήξη συνεδρίαση. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί 9 με τους συντονιστές και 10 η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.